Συνάδελφοι, δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε. Οι πράσινοι εκπροσωπούνται, κάποιοι σοσιαλιστές είναι εδώ. τι άμα συνεχίσουμε έτσι Λοιπόν, αρχίζουμε σημείο 11 Ταμείο αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ρώσα Εστερά Φραγκούτε, η συγγήτρια έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το Ταμείο Συνοχής δημιουργήθηκε το 2002, όπως γνωρίζετε. Είναι το ε, μέσο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ανταποκρίνεται σε καταστροφές που λαμβάνουν χώρα σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Εφαρμόζεται και στα κράτη-μέλη και στις πένταξη χώρες και στις χώρες που χωρίς να είναι μέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχουν ε, προβλεφθεί να είναι δικαιούχες. Ε, παλιότερα δεν υπήρχε κανένα τέτοιο μέσο για περιπτώσεις καταστροφής και θεομηνίας. Νομίζω ότι είναι ένα μέσο πάρα πολύ σημαντικό, πολύ χρήσιμο ε, όλα τα τελευταία χρόνια. Το 2005 προτάθηκε μια τροποποίηση γιατί είχαν εμφανιστεί δυσκολίες στην εφαρμογή του, αλλά τελικά το Συμβούλιο απέρριψε αυτές τις αλλαγές γιατί προτείνονταν αλλαγές στα κόστη και στα κριτήρια οπότε τις απέρριψε το Συμβούλιο. Στη νέα φάση Πέρσι το 2012 υποβάλαμε μια έκθεση δική μου για να δούμε πώς θα έπρεπε να τροποποιηθεί ο κανονισμός του Ταμείου Συνοχής με, έτσι ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικός. Και βέβαια διορθώναμε τα λάθη τα οποία είχαμε εντοπίσει τα τελευταία χρόνια. Ποιες είναι οι αλλαγές προτείνουμε και σε τι διαφωνούμε με την Κομισιόν. Καταρχήν, ε, τι είναι οι σημαντικές ε, τεράστιες περιφερειακές καταστροφές. Ε, ε, το διατηρούμε, 3 δισεκατομμύρια ευρώ, πάνω από αυτό το ποσό θεωρείται τεράστια η περιφερειακή καταστροφή. Όμως, τα δύο τρίτα τομεία προβλεπόντουσαν για περιφερειακές καταστροφές. Ο κανονισμός λέει συγκεκριμένα ότι είναι επιλέξιμες οι καταστροφές που ε, επηρεάζουν την πλειοψηφία του πληθυσμού ή που επηρεάζουν τις συνθήκες ε, οικονομικής ζωής, την οικονομική σταθερότητα ε, και έχουν σημαντικές επιπτώσεις επί αυτών. Είναι λίγο ασαφής ε, και αόριστη αυτή η διατύπωση και πολλές ε, περιφέρειες ε, είχαν κάποιες προσδοκίες, έφταναν τα ντοσιά του στην Κομισιόν και η Κομισιόν πολλά τα απέριπτε. Οπότε απογοητεύονταν οι περιοχές, οι περιφέρειες αυτές. Προτείνουμε αλλαγή και η Κομισιόν το πρότεινε άλλωστε και εμείς. Οπότε λέμε <clears throat> πλέον προτείνουμε όταν φτάνουμε στο 1% του περιφερειακού ΑΕΠ στις περιοχές ΝΟΤΣ 2, ΝΑΤΣ 2, να είναι επιλέξιμες. Πολύ συγκεκριμένο ε, ποσοτικό κριτήριο. Η Κομισιόν προτείνει 1,5%. Εγώ θα προτείνω 1%. Η Επιτροπή των Περιφερειών επίσης προτείνει 1%. Εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε, υποβάλλετε τροπολογίες. Άλλο ζήτημα σημαντικό ήταν οι προκαταβολές. Σε περίπτωση καταστροφής τέτοιου τύπου είναι πολύ σημαντικό να γίνονται αμέσως πληρωμές έτσι ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Η Κομισιόν προτείνει ε, το 10% των ποσού να μπορεί να δοθεί ως προκαταβολή με ανώτατο όριο τα 30 εκατομμύρια. Το δέχομαι και εγώ και το προτείνω. Αυτό επιτρέπει άμεση και μεγαλύτερη παρουσία. Ε, με βοήθεια. Απλοποιείται επίσης η διαδικασία. με άμεσες ε, πληρωμές, γρήγορες πληρωμές. Μετά ε, κατέθηκαν και διάφορα άλλα αιτήματα για καταστροφές βραδίας εξέλιξης όπως η ξηρασία. Ε, και η Επιτροπή των Περιφερειών προτείνει να τις περιλάβουμε Μάλιστα περιλαμβάνει και τις πλημμύρες θα δούμε αν θα, το, αν θα τις συμπεριλάβουμε και εμείς. Δεν ξέρω αν οι πλημμύρες είναι καταστροφές βραδιάς εξέλιξης. Ο κανονισμός μέχρι τώρα έλεγε μέχρι, από τη στιγμή που λαμβάνει χώρα η καταστροφή μπορεί να περάσουν μέχρι 10 εβδομάδες για να ζητήσει κανείς η περιφέρεια, δηλαδή βοήθεια. Ε, διευρύνουμε αυτή την ε, προθεσμία. 10 ε, εβδομάδες είναι λίγο μικρό χρονικό διάστημα γιατί το πιο σημαντικό εκείνη την εποχή είναι ε, να λυθούν τα άμεσα και επίγοντα προβλήματα ε, οπότε δεν είναι εύκολο ε, να υποβληθεί η αίτηση στο αίτημα στις 10 εβδομάδες γι' αυτό και διευρύνουμε αυτή την προθεσμία. Μετά, για για ποια πράγματα μπορεί να ζητηθεί βοήθεια. Υπάρχει ένα κεφάλαιο που αφορά τις ε, υποδομές και η Επιτροπή των Περιφερειών ε, προτείνει ε, στο πλαίσιο αυτό των υποδομών να συμπεριλαμβάνεται όχι μόνο η επισκευή των υποδομών αλλά και η μεταφορά τους έτσι ώστε ενδεχομένως να αποφευχθεί η επανάληψη της καταστροφής σε παρόμοιο φαινόμενο. Τι άλλο. Μερικές φορές οι καταστροφές γίνονται σε διασυνοριακές περιοχές που δεν ειναι νατς NATS2. Ε, λέμε παρόλο ότι δεν ειναι νατς NATS2, σε αυτή την περίπτωση επειδή είναι διαμεθοριακές οι καταστροφές να μπορούν να είναι δικαιούχες βοήθειας. Μετά η Επιτροπή των Περιφερειών λέει και το εξή που μου φαίνεται ενδιαφέρον. Οι νατς 2 ε, θα πρέπει να ζητούν τη βοήθεια, αλλά ενδεχομένως η καταστροφή να έχει επηρεάσει μικρότερες ζώνες που δεν ειναι νατς NATS2 και παρόλα αυτά το σύνολο αυτών των μικρών περιοχών να δίνει ένα πληθυσμό ίδιο με αυτόν προβλέπει να ΝΑΤΣ2 οπότε σε αυτήν την περίπτωση να μπορούν να ζητούν βοήθεια. Μετά, ε, για την προθεσμία εκτέλεσης ε, ήταν ένα έτος, ε, εμείς το αυξάνουμε κατά έξι μήνες, μισή χρόνο, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, να απορροφηθούν δηλαδή τα κονδύλια. Και κάτι άλλο το οποίο δεν το προτείνει η Κομισιόν αλλά θεωρούμε ότι είναι σημαντικό, είναι τεχνικό θέμα, οι περιφερειακές καταστροφές συνήθως πλήττουν ε, περιφέρειες που έτσι κι αλλιώς αντιμετωπίζουν προβλήματα. Για παράδειγμα, η περιοχή της Λόρκα ή της Σαρδινίας, θυμάμαι τελευταία, είναι μικρές περιφέρεις με περιορισμένους πόρους και περιορισμένες υποδομές. Οπότε ένα τμήμα του ταμείου, 2% προτείνουμε, όπως και η Επιτροπή των Περιφερειών, να μπορεί να χρησιμοποιείται για τεχνική συνδρομή. Ε, για να γίνουν τα, τα σχέδια, οι μελέτες, ε, οι αρχιτεκτονικές και άλλες που χρειάζονται. Αυτά. Ε, ο χρόνος πιέζει αλλά νομίζω μπορούμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Ε, τη Δευτέρα θα είναι έτοιμη η έκθεση για να γίνει μετάφραση και αν τηρηθούν οι προθεσμίες του χρονοδιαγράμματος ε, είναι δυνατό η ψηφοφορία να γίνει φέτος το Γενάρη μάλλον το 2014 και να πάει στην Ολομέλεια το Μάρτιο. Μετά βέβαια έχουμε τον τριμερή διάλογο αλλά νομίζω ότι αν δεν επηρεάσουμε τον προϋπολογισμό, όλα τα υπόλοιπα μπορούν εύκολα να συμφωνηθούν. Ε, βέβαια, στις δημοσιονομικές προοπτικές το, ταμείο, το προπολογισμό ταμείου μειώθηκε από το 1 δισεκατομμύριο στα 500 εκατομμύρια. Ε, Παρ' όλα αυτά, οι καταστροφές αντί να μειώνονται, αυξάνονται. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να παραμείνουμε περιορισμένοι σε αυτό το πλαίσιο και να διορθώσουμε ό,τι μπορούμε να διορθώσουμε. Ευχαριστώ. Uh, λοιπόν, ευχαριστούμε Ρόζα Σκιώδης. Μόνο ο Νίκος Χρυσόγελος βρίσκεται εδώ από τους Σκιώδης. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Α, και εσείς θα μιλήσετε για τους σοσιαλιστές. Ο Νίκος, έχετε το λόγο. Ε, νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση για να επανανεργοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ελεγγύης είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, ιδιαίτερα σε μια εποχή που αυξάνονται οι φυσικές καταστροφές. Βλέπουμε παντού ότι η κλιματική αλλαγή ε, αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση ακραίων καιρικών φαινομένων και βλέπουμε να υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις σε διάφορες περιφέρειες. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι λόγοι όπως η ξηρασία, οι πλημμύρες, ε, οι μεγάλες πυρκαγιές. Ε, νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί σύντομα μια ε, συμφωνία με το Συμβούλιο έτσι ώστε πραγματικά να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην ε, χρήση του Ταμείου. Συμφωνούμε σε πολλά από αυτά που η συγγήτρια ε, παρουσίασε. Θα δούμε και την έκθεση. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει συνεργασία. Μία σημαντική διάσταση την οποία είχαμε τονίσει και στην έκθεση που έγινε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι ότι πρέπει να προβλέπεται και η αποτροπή επανάληψη των ίδιων φαινομένων. Δηλαδή, όταν γίνεται αποκατάσταση, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ε, η αξιολόγηση των, ε, της εμπειρίας από την καταστροφή, τι συνέβαλε στη μεγιστοποίηση μιας καταστροφής, έτσι ώστε τα έργα που θα γίνουν, οι παρεμβάσεις που θα γίνουν, να αποτρέπουν την επανάληψη. Πολλές φορές βλέπουμε να επαλαμβάνονται τα ίδια φαινόμενα πλημμύρας, γιατί υπάρχουν προβλήματα στις υποδομές, για παράδειγμα ένας, ε, ένα μπαζωμένο ρέμα, ένα ποτάμι το οποίο έχει κλείσει ή κακή ε, διαστασιολόγηση των γεφυρών μπορεί να οδηγήσει σε πλημμύρες. Αλλά αν δεν αποκατασταθεί αυτό το πρόβλημα μπορεί αυτό να επαλαμβάνεται δύο και τρεις φορές όπως έχουμε δει σε πολλές περιοχές. Νομίζω κάθε φυσική καταστροφή θα πρέπει να μελετάτε να αξιολογούνται τα αίτια που οδήγησαν στην ένταση του φαινομένου. Πολλές φορές έχουμε ένα συνδυασμό ε, φυσικών φαινομένων αλλά και ε, λάθος κατασκευών ή λάθος επιλογών στο πεδίο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη μέσα στο σχέδιο για την αποκατάσταση και μία έκθεση συμπερασμάτων για το πού οφείλεται η έκθεση καταστροφή. Νομίζω θα είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν είναι λογικό να, να δαπανάμε συνέχεια δημόσια χρήματα για λάθος ε, επιλογές ή λάθο κατασκευέ έργων. Ε, νομίζω ότι πρέπει να εντάξουμε και τα θέματα και τη ξηρασία και των πλημμυρών ε, στους στόχους. Είναι και βραδία εξέλιξη, αλλά βέβαια, όπω είπαμε, συνδέεται και πολλέ φορέ με κατασκευαστικά θέματα, τουλάχιστον οι πλημμύρε ή με κακή διαχείριση των δατικών πόρων πρέπει να συνδέουμε αυτά τα θέματα γιατί υπάρχει και σχετική νομοθεσία, αλλά πρέπει να τα συνδέουμε και με τη διαχείριση επίπεδο υδρολογικής λεκάνης, δηλαδή παράδειγμα όταν συμβεί κάπου μία πλημμύρα και οι αρχές να εξετάζουν κατά πόσον όλο αυτό το, όλη αυτή η ζημιά, η καταστροφή, οφείλεται και σε κακή διαχείριση των εντατικών πόρων. Είτε αυτό είναι ποτάμια που είναι διασυνοριακά, είτε ποτάμια που είναι σε μια περιφέρεια αλλά πολλές φορές πάνε προβλήματα και μέσα στον αστικό χώρο από κακή διαχείριση ε, των υδάτων. Ε, νομίζουμε ότι είναι σωστό ε, να ε, αυξηθεί και να το όριο για την καταβολή κάποιας βοήθειας από το 1% του περιφερειακού έψη στο 1,5% και να υπάρξει μεγαλύτερος χρόνος για αποκατάσταση, δηλαδή να έχουμε 16-18 μήνες, γιατί πράγματι μερικές φορές η, η όλη διαδικασία είναι πάρα πολύ χρονοβόρος. Δηλαδή μέχρι να γίνουν τα σχέδια, οι μελέτες, να γίνουν τα έργα, να προκυριθούν κτλ. Η εμπειρία δείχνει ότι σε πολλές χώρες αυτό είναι μια δικασία πολύ επίπονη και γραφειοκρατική. Ε, άρα θα πρέπει να αυξηθεί ίσως σε 1,5 χρόνο η προθεσμία εκτέλεση των έργων. Και επίσης και ο χρόνος που χρειάζεται μία αρχή να υποβάλει την έκθεση. Ε, οι δέκα εβδομάδες ίσως είναι πολύ λίγες γιατί εκείνη τη στιγμή υπάρχει η επικέντρωση κυρίως στο πώς θα βοηθεί ο πληθυσμός ή πώς θα γίνουν κάποιες ενέργειες. Άρα πράγματι συμφωνούμε να αυξηθεί ο χρόνος μέσα στον οποίο μία αρχή θα μπορεί να υποβάλει έτσι για το ε, ταμείο. Α, και, και ένα τελευταίο. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένα δίκτυο ειδικών που θα βοηθάνε περιφέρειες να υποβάλουν φακέλους. Ε, πολλές φορές αυτοί που πλήττονται είναι, όπως είπε και η συγγήτρια, περιφέρειες που έχουν μικρές δυνατότητες, έχουν περιορισμένες δυνατότητες και δεν είναι σε θέση να προετοιμάσουν εκθέσεις, σχέδια κτλ. Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία λίστα, μία βάση δεδομένων όπου θα μπορεί να υπάρχει ανταλλαγή εμπειριών και αλληλοβοήθεια για να υποβάλλονται ε, σωστά σχέδια και να μην απορρίπτονται λόγω ανεπάρκειάς τους. Thank you. Um, Ευχαριστούμε. Η Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να χαιρετήσω ολόθερμα την πρόταση αυτή για την ε, μεταρρύθμιση του Ταμείου Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι η πρόταση κινείται στην σωστή κατεύθυνση. Από το 2005 είδαμε ότι οι περιφέρειες περιμένουν και πάρα πολλές περιμένουν σημαντικότατες και γρήγορες ε, βοήθειες ε, για να αντιμετωπίσουν τις φυσικές καταστροφές. Πρέπει λοιπόν να πλουστευτούν διαδικασίες και έχουν περάσει 8 χρόνια όπου αντιτίθεται το Συμβούλιο. Θεωρώ ότι είναι δραματικό και πραγματικά ας μην ξεχνάμε ότι μια σημαντικότατη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ελεγγύη. Ο Επίτροπος Χάν πρόσφατα είπε ότι θα έχουμε 400 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ελληνική στην Τσεχία, τη Ρουμανία καθώς επίσης και σε άλλες χώρες που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Εμείς όντως εγκρίναμε αυτά τα 400 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον στον διορθωτικό προπολογισμό που εγκρίναμε στην προηγούμενη ολομέλεια της, του Στρασβούργου. Βέβαια πρέπει να αναθεωρηθεί ο καονισμός αυτός για το Ταμείο Λιλεγγύης. Θα πρέπει τα χρήματα αυτά να δοθούν πολύ γρήγορα και σε άλλες χώρες όπως η Ιταλία που χρειάστηκε να περιμένει πάρα πολύ καιρό προκειμένου τη δοθεί απαραίτητη χρηματοδότηση. Η μεταρρύθμιση αυτή λοιπόν αυτή η επίγη είναι πιο εύκολο τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί σε μια καταστροφή σε μια, στην άλλη γωνιά του κόσμου από ότι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο. Το Ταμείο Λιλεγγύης ε, επενδύει πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε 56 περίπου περιπτώσεις από τότε που δημιουργήθηκε το 2002. Ξέρουμε όμως ότι επιτόπου έχουμε πάρα πολλές φυσικές καταστροφές, πολύ περισσότερες από τον αριθμό που ανέφερα και αναφέρομαι βέβαια και στις ανθρωπογενείς καταστροφές που υπερβαίνουν από το 2002 τον αριθμό που παρέθεσα πριν από λίγο. Οι συναδελφοί μου το είπανε ότι βλέπουμε όλο και περισσότερο τις καταστροφές αυτές να αυξάνονται λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη και των κλιματικών αλλαγών. Πρέπει λοιπόν και τη συνιστός αυτή να την συμπεριλάβουμε στην ανάλυση που κάνουμε. Και ξέρετε ότι για πολλές καταστροφές δεν μπορέσαμε να δώσουμε κάποια βοήθεια υποστήριξη. Για παράδειγμα στη δική μου περιφέρεια τον Ιούνιο στην νότιο-δυτική Γαλλία είχαμε φυσικές καταστροφές που στήχησαν τη ζωή σε πολλού ανθρώπου, καθώ επίση και πολλέ καταστροφέ και ζημιές που φτάνουν εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε ότι ε, σε ορισμένες πόλεις της νοτιωτικής Γαλλίας ε, ε, υπάρχουν πάρα πολλά μνημεία τα οποία καταστράφηκαν. Στην Λούρδη, για παράδειγμα, ξέρετε ότι υπήρχαν πολύ σημαντικότητες πλημμύρες και σημαντικότητες καταστροφές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ποια είναι τα κριτήρια τα οποία είναι ασαφή αυτή τη στιγμή όσον αφορά τι φυσικέ καταστροφέ και πολύ φοβάμαι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύγχυση που έχει να κάνει και με την γαλλική γραφειοκρατία. Θα ήθελα λοιπόν να καταφέρουμε να προχωρήσουν περισσότερο με τις προτάσεις αυτές, με το 10% καθώς επίσης και με το 1,5% όσον αφορά το περιφερειακό ΑΕΠ. Πρέπει το ταμείο αυτό να είναι απλό, χρειαζόμαστε ένα υψηλό βαθμό διαφάνειας και μια πλούστευση του συστήματος στις συζητήσεις επίσης ε, που γίνονται και είναι πάρα πολύ σημαντικό εν ώψη των ευρωπαϊκών εκλογών να δείξουμε ότι μπορούμε γρήγορα και αποτελεσματικά να αποκριθούμε στις ανάγκες των ε, περιφερειών μας. Δεν νομίζω πάλι ότι ε, Πρέπει, μάλλον, πρέπει να λάβουμε υπόψη μα και τον διαφορετικό στελεστή όσον αφορά το ΑΕΠ των περιφερειών. Ενδεχομένω κάποιε περιφέρειες να χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη από κάποιε άλλε. Υποστηρίζω επίση την πρόταση τη κυρία Εστάρα να παραταθεί η περίοδο τη προθεσμία προβλέπει, η χρονική περίοδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να τονίσουμε την ιδέα της αλληλεγγύης σας, μη μειώνουμε τα ποσά όπως, προτάθηκε από το Συμβούλιο, ακριβώς επειδή δεν είχε χρησιμοποιηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, μα δεν είχε χρησιμοποιηθεί το ταμείο αυτό ακριβώς επειδή το Συμβούλιο είχε αντιταχθεί στη χρήση του, είχε μπλοκάρει τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη από το ταμείο αυτό. Αν μειωθεί λοιπόν η χρηματοδότηση του ταμείου αυτού, θα πρέπει να ψάξουμε αλλού τους πόρους, ενδεχομένως από τα διαφορετικά ταμεία, προκειμένου να καταφέρουμε μη άλλο να έχουμε ένα σύστημα πρόληψης των καταστροφών ή μια καλύτερη διαχείριση των φραγμάτων ή των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών που ενδεχομένω να παρουσιάζουν μεγαλύτερε κινδύνου ε, για φυσικέ καταστροφέ. Α μην ξεχνάμε όμω ότι ε, και στα πλαίσια του Interreg θα πρέπει να δοθεί απαραίτητη χρηματοδότηση. Οι φυσικέ καταστροφέ δεν γνωρίζουν σύνορα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε υψηλότερο επίπεδο ελεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριο Σταυρακάκη έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την παρουσίαση και την τοποθέτηση που μας έκανε. Όπως ίσως να γνωρίζετε, είμαι ο εισηγητής της γνωμοδότησης τη Επιτροπής Προπολογισμών και χθε είχαμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων όπου παρουσίασα το σχέδιο γνωμοδότησής μου περιορίζοντάς το σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας της ε, Μπάλης. Καλωσόρισα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Σε ορισμένα θέματα όμω, κάλεσα την Επιτροπή Προπολογισμών να πάει ένα βήμα περαιτέρω. Υποστήριξα το κριτήριο για την κινητοποίηση του Ταμείου Ελληνική για τι λεγόμενε έκτακτε περιφερειακέ καταστροφέ. Ωστόσο, πρότεινα το κατώτατο όριο τη ενεργοποίηση να τεθεί στο 1% του, 1 του περιφερειακού ΑΕΠ αντί του 1,5%. Υποστήριξα τη δυνατότητα να γίνονται προκαταβολέ κατόπιν ετήσεω τη πληγή τη χώρα και πρότεινα να τεθεί το ανώτατο όριο των προκαταβολών στο 15% του αναμενόμενου ποσού τη οικονομική ενίσχυση, που δεν θα υπερβαίνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ καθώ δεν έχει καμία δημοσιονομική επίπτωση. Ωστόσο επέστησα την προσοχή στο ότι η πρόταση τη Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 4α παράγραφος 3 για τη χρηματοδότηση των προκαταβολών ως έχει προποθέτει αλλαγή του κανονισμού των κοινών διατάξεων του CPR, το οποίο είναι προβληματικό στην παρούσα φάση και μόλι την περασμένη εβδομάδα ψηφίστηκε και γι' αυτό θα πρέπει να αναζητήσουμε εναλλακτικού τρόπου χρηματοδότησή του. Επιπλέον πρότεινα να επεκταθεί το χρονικό διάστημα δυνατότητα χρήση τη ενίσχυση του Ταμείου από 12 στου 18 μήνε, καθώ η νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων, για παράδειγμα, σε πολλέ χώρε είναι αρκετά χρονοβόρα. Η πρόληψη των καταστροφών, αγαπητοί συνάδελφοι, αποτελεί ύψιστη σημασία. Γι' αυτό και το Ταμείο θα πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τα άλλα χρηματοδοτικά μέσα, όπως τα ευρωπαϊκά διαθροτικά και υπηρετικά ταμεία, ώστε να μπορέσουν να επιτευχθούν συνέργειες. Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε και η πρότασή μου στην Επιτροπή Προπολογισμών να καταστεί τεχνητή βοήθεια επιλέξιμη δαπάνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Um, Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο κύριος Βλάσεκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη γνωμοδότηση. Είναι υψηλής ποιότητας το κείμενό της και ίσως πρέπει να προβληματιστούμε για κάποια θέματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται στις περιφέρειες ΝΑΤΣ 2 και προβλέπει 1,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, αλλά δεν περιορίζονται σε διοικητικές περιφέρειες πολλές φορές οι καταστροφές, πολλές φορές είναι διασυνοριακά τα φαινόμενα. Γι' αυτό λοιπόν θα έπρεπε να καλύπτεται μεγαλύτερη επιφάνεια και να χρησιμοποιείται αυτή ως βάση για τον υπολογισμό του κριτηρίου του εγχωρίου προϊόντος. Δεν νομίζω ότι πρέπει να έχουμε σε σημείο εκκινήσεως μόνο τις περιφέρειες ΝΑΤΣ 2. Αυτό το 1,5% ΑΕΠ δεν αρκεί αν αναλογιστούμε τις πιο σημαντικές καταστροφές, έκρηξη της έτνας, πλημμύρες, περιπτώσεις όπου δύσκολα θα αξιολογηθούν οι επιπτώσεις με βάση αυτά τα κριτήρια. Χρειάζονται λοιπόν προσαρμογές και τα, οι τιμές αναφοράς πρέπει να μειωθούν. Εγώ θα έλεγα 1% του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος. Εκτός αυτού πρέπει να απλουστευτούν οι διοικητικές διαδικασίες, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζεται να ενημερώνονται και οι ενδιαφερόμενοι. Αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο. Οι δε αιτήσει θα πρέπει να μπορούν να ε, τίθενται, να υποβάλλονται και μετά από παρέλευση 10 εβδομάδων. Τέτοιες καταστροφές πρέπει να παρακολουθούνται για μακρότερα χρονικά διαστήματα για να έχουμε μία ιδέα σχετικά με το εύρος των επιπτώσεων που έχουν και συχνά περνάει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι να κηρυχθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να αξιολογηθούν οι ζημίες. Ιωάννης, ε, Ε, πριν σου δώσω το λόγο θα ήθελα να σε ρωτήσω αν μπορείς να μας ενημερώσεις τι ξέρουμε για τη θέση του Συμβουλίου σήμερα. Γιατί έγιναν διαβουλεύσεις στο παραδοσιακό επίπεδο. Ε, ε και, ε, ποια είναι η επίσημη θέση των Υπουργών Οικονομικών. Και υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το Συμβούλιο, γιατί το δικό μας χρονοδιάγραμμα είναι αισιόδοξο και θέλουμε ε, το αργότερο τον Απρίλιο να ψηφιστεί στην Ολομέλεια η γνωμοδότηση. Πες μας λοιπόν ενημέρωσέ μας τι γνωρίζεις, που βρίσκονται τα πράγματα και αν υπάρχει κάποια πληροφορία σχετικά με την έκθεση πρωτοβουλίας και πόσο χρησιμοποιήσαμε, τι ποσό χρησιμοποιήσαμε σε αιτήσιο ε, επίπεδο. νομίζω μόνο για τη Γερμανία είχαν ετηθεί 400 εκατομμύρια. Δηλαδή πώς ε, αποφάσισαν από το 1 εκατομμύριο να κατέβουν στα 500 εκατομμύρια. Ενώ οι αιτήση είναι για περισσότερα ποσά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να αρχίσω με τα θέματα που θέσατε εσείς για το Συμβούλιο. Ακόμα δεν έγινε συνάντηση με το Συμβούλιο για να συζητηθεί η πρόταση της Κομισιόν. Η πρώτη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για Διαρθρωτικές Δράσεις προγραμματίζεται για το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Υπάρχει προσωρινό χρονοδιάγραμμα και για κάποιες άλλες συνεδριάσεις μέσα στο πρώτο τρίμηνο του επομένου έτους, αλλά αυτό είναι προσωρινό και δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο, θα, γρήγορα θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εξαρτάται και από τη θέση που θα λάβουν τα κράτη-μέλη επί των διαφόρων ε, θεμάτων που προτείνουμε. Δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πρόοδο που θα υπάρξει στο Συμβούλιο. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω και κάτι ακόμα, το Συμβούλιο δεν ε, καίγεται να προχωρήσει γρήγορα γιατί ο κανονισμός ε, για το Ταμείο Αλληλεγγύης στο τωρινό υπάρχει και δεν λύγει. Οπότε από αυτή την πλευρά δεν υπάρχει άμεση πίεση στο Συμβούλιο. Βέβαια, σε πολιτικό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να επιτελεστεί πρόοδο σε αυτό το θέμα και να ε, θεσπιστεί, να εγκριθεί ο κανονισμός πριν ε, τελειώσει η θητεία αυτού του Κοινοβουλίου πριν από τις ευρωεκλογέ. Τώρα, η ετήσια ανάλωση του Ταμείου. Από το 2002 είχαμε ένα δις ευρώ ως μέγιστο διαθέσιμο ποσό πέρα από τον κατακτικό ε, προϋπολογισμό αυτό το ένα δις δεν ήταν ποτέ στόχος δαπανών αλλά υπήρχε μια κατανομή που δηλαδή, ε, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο χειρότερο σενάριο. Ο κανονισμός καθ' αυτός δεν προβλέπει λεπτομέρειες σχετικά με την χρήση αυτών των κονδυλίων. Λέει ότι το Ταμείο ή τα κονδύλια ε, που περιέχει θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με τρόπο ε, σόφρονα για να μην εξαντληθούν τα κονδύλια του Ταμείου πριν από την παρέλευση ενός έτους πρέπει να διατηρηθούν μέχρι το τελευταίο τρίμηνο κάθε χρόνο και πρέπει να υπάρχουν προβλέψεις ώστε αν σε πολύ κακή χρονιά έχουμε το σεισμό στη Λάκουλα και την πλημμύρα στη, πλημμύρα στη Γερμανία και πυρκαγιές στην Ισπανία, όλες οι καταστροφές μέσα σε ένα χρόνο, παρόλα αυτά να μπορούμε να καλύπτουμε τις ανάγκες με τα κονδυλία που διαθέτουμε. Η χρήση του Ταμείου έχει παρουσιάσει μεγάλες διακυμάνσεις τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρξαν χρόνια όπου χρησιμοποίησαμε 100 εκατομμύρια και ούτε καν, άλλες φορές χρησιμοποίησαμε, δώσαμε πάνω από 800 εκατομμύρια. Αυτό είναι απρόβλεπτο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2002, όταν δημιουργήθηκε το Ταμείο, επεξεργάστηκε μία μέθοδο υπολογισμού των επιχορηγήσεων με βάση την αρχή ότι δεν πρέπει να υπάρχει ε, το στοιχείο του με τη σειρά προτεραιότητος αλλά θα εξετάζονται οι καταστροφές στην πορεία του έτους και τα κράτη-μέλη τα πιο φτωχά παίρνουν περισσότερα ποσά αν χρειαστούν από ό,τι τα πλουσιότερα κράτη-μέλη. Και το ένα δις θα πρέπει να υπαρκεί για να γίνονται όλα αυτά. Ξέρετε τη μέθοδο στην οποία καταλήξαμε και η οποία απέδειξε ότι μπορούμε να χειριστούμε τις καταστροφές και η μέθοδος υπολογισμού όντως ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και ποτέ δεν εξαντλήσαμε τα κονδύλια του Ταμείου. Κατά μέσον όρο χρησιμοποιήσαμε το Ταμείο τα προηγούμενα 11 χρόνια κατά το 1 τρίτο σε αιτήσια βάση. Αλλά όπως σας είπα κάποιες φορές δίναμε περισσότερα, άλλες φορές λιγότερα. Τώρα, ε, αναφέρομαι σε αυτά που είπε η συγγήτρια και διάφορα μέλη της Επιτροπής. Το σκεπτικό της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ουσιαστικά να βελτιωθεί η λειτουργία του υφισταμένου Ταμείου Αλληλεγγύης για να ανταποκρίνεται πιο ταχαίως, με απλούστερο τρόπο, να είναι πιο εύχριστο, να είναι σαφέστερες οι διατάξεις του. Θεωρήσαμε ότι θα ήταν σημαντικό όμως να διατηρήσουμε την το, το σκεπτικό του ίδιου του Ταμείου, ε, το ιδρυτικό του σκεπτικό και οι προτάσεις μας δεν θα έπρεπε να αυξήσουν τις δαπάνες μεταξύ άλλων διότι με το, στα πλαίσια του παρόντος κλίματος τα κράτη-μέλη δεν είναι πιθανό να δεχτούν προτάσεις που θα σημάνουν αύξηση των δαπανών. Και πάλι εδώ το υπόβαθρο είναι ότι στα πλαίσια του νέου πολιετούς δημοσιονομικού αυξήθηκε κατά 50% το ταμείο, αλλά αυτό δεν βοηθάει όταν πρόκειται να προσθέσουμε κι άλλα στοιχεία στο υφιστάμενο ταμείο. Τώρα, ένα θέμα είναι ότι θέλουμε απλούστερα κριτήρια ή ένα απλό ενιαίο κριτήριο για τις περιφερειακές καταστροφές που μάλλον είναι η εξαίρεση από τον κανόνα. Ο κανόνας είναι μεγάλες καταστροφές, αλλά ο κανονισμός προβλέπει κινητοποίηση του Ταμείου και για περιφερειακές μικρότερες καταστροφές. Ε, αναφέρθηκε προηγουμένως το κριτήριο που έχουμε στον παρόντα κανονισμό και είπαμε ότι είναι περίπλοκα και θέλουμε να τα αντικαταστήσουμε με ένα απλό κριτήριο με βάση το ΑΕΠ. Εμείς είπαμε 1,5%. Η πρόταση εδώ που ακούστηκε είναι 1%. Το 1,5% που προτείνουμε εμείς το εξετάσαμε πολύ προσεκτικά και προτείνουμε αυτό το ποσοστό ακριβώς διότι θα οδηγήσει σε κινητοποίηση του Ταμείου για περιφερειακές καταστροφές που ανταποκρίνονται στην πρακτική του παρελθόντος. Εάν μειώσουμε το κατόφλι στο 1% του ΑΕΠ θα συμπεριλαμβάνουμε στο μέλλον έναν αριθμό μικρότερων καταστροφών που τώρα δεν είναι πιθανόν να χαρακτηριστούν επιλέξιμες, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των κινητοποιήσεων και δαπανών. Και δεν είμαι απόλυτα βέβαιος ότι η μείωση του κατοφλίου στα 1% θα αποστείλει το σωστό μήνυμα σήμερα. Τα... Οι προκαταβολές που προτείνουμε είναι πολύ σημαντικές γιατί μας επιτρέπουν ταχύτερη παρουσία από ό,τι συμβαίνει σήμερα ταχύτερη ανταπόκριση. Τώρα, αν περιορίζονται στο 10% ε, κατά μέγιστον 30 εκατομμύρια και 15% 40 εκατομμύρια όπως προτάθηκε, αυτό δεν νομίζω ότι ε, έχει ουσιώδη διαφορά. Η Κομισιόν δεν αντιτίθεται σε μια τέτοια πρόταση. Όμως το ερώτημα είναι αυτοί οι πόροι από πού θα αντληθούν. Εδώ χρειάζεται περαιτέρω προβληματισμός και συζητήσαμε και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών το θέμα χθε και είπαμε ότι θα αναζητήσουμε εναλλακτικέ στις τωρινές προτάσεις που πράγματι θα απαιτήσουν τροποποίηση του κανονισμού των κοινών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία που τώρα εγκρίθηκε και δεν είναι το καλύτερο αυτό. Αν υπάρχουν εναλλακτικέ άλλες η Κομισιόν δεν θα διαφωνήσει αν είναι βιώσιμες βέβαια. Τώρα, οι 10 εβδομάδες περίοδος ε, υποβολής αιτήσεων που αναφέρθηκε και κάποιοι ομιλητέ είπαν ότι είναι πολύ σύντομη περίοδος. Οι 10 εβδομάδες είναι μια πρόταση η οποία αναφέρεται στον ε, τωρινό κανονισμό, αυτό δεν το τροποποιούμε. Και αυτές οι δέκα εβδομάδες επιχειρούν να βρουν μια ισορροπία μεταξύ της ταχείας ανταπόκρισης σχετικά και και της παροχής μιας περίοδου κατάλληλης ώστε το κράτος μέλος να αξιολογήσει τη ζημιά. Πολλές φορές ξέρουμε ότι κάνουν την αίτηση στα κράτη-μέλη την τελευταία στιγμή, οπότε είναι μικρή. Το αν όμως πρέπει να παρατείνουμε αυτή την προθεσμία δεν ξέρω αν είναι τόσο καλή ιδέα, γιατί η ιδέα είναι να ανταποκρίνεται πιο γρήγορα το Ταμείο. Αν παρατείνουμε την ε, περίοδο υποβολή, υποβολής αιτήσεων στις 12 ή 15 εβδομάδες, θα καθυστερεί να κινητοποιηθεί το Ταμείο και θα μας επικρίνουν μετά γι' αυτό κάτω από συγκεκριμένες και ειδικέ συνθήκες όπου μια καταστροφή συνεχίζεται για μακρότερο χρονικό διάστημα, πάντα ήταν δυνατόν και θα συνεχίσει να είναι δυνατόν να προστίθενται πληροφορίες λεπτομερέστερες σε ένα μετέπειτα στάδιο και μετά την υποβολή της αίτησης. Αναφέρθηκε ότι το, η περιφέρεια ΝΑΤΣ 2 ίσως δεν είναι κατάλληλη αναφορά, κατάλληλο σημείο αναφοράς για τις καταστροφές. Πρέπει να καθορίσουμε τις καταστροφές σε σχέση με κάτι και σε σχέση με κάτι για το οποίο διαθέτουμε στατιστικά στοιχεία. Αν οι καταστροφές δεν ε, περιορίζονται σε διοικητικές περιφέρειες και διευρύνονται, τότε μπορούμε να συμπεριλάβουμε περισσότερες περιοχές ΝΑΤΣ 2. Και σε αυτή την περίπτωση ο σταθμισμένος μέσος όρος του ΑΕΠ αυτών των δύο ή τριών περιοχών θα λαμβάνεται υπόψη ως σημείο αναφοράς. Τώρα, για διασυνοριακές περιοχές. Αυτό ε, δημιουργεί μια δυσκολία. Δηλαδή, όπως είναι φτιαγμένο το Ταμείο, ε, αναφέρεται στα κράτη-μέλη. Δηλαδή, πάει να βοηθήσει τα κράτη-μέλη. Να τα βοηθήσει να επομιστούν το οικονομικό βάρος μιας καταστροφής. Αν δούμε τις διασυνοριακές περιοχές, είναι δύσκολο να πούμε σε σχέση με ποια χώρα πρέπει να κινητοποιηθεί το Ταμείο, αν θεωρηθεί μια ενιαία καταστροφή. Μία και μόνο. Μπορεί να είναι δυνατόν να κινητοποιηθεί για δύο χώρες αν έχει διασυνοριακές επιπτώσεις η καταστροφή ή και διατηρούμε την πρόταση. Αν σε ένα κράτος μέλος υπάρχει σοβαρή καταστροφή, ένα γειτονικό κράτος μέλος πάντα μπορεί να υποβάλει αίτηση χωρίς να πληρεί το κατόφλιο και η διάταξη διατηρείται, η πρόβλεψη διατηρείται. Τώρα, ε, περίοδος εφαρμογής ε, που θα επεκταθεί στους 18 μήνες. Αυτό δεν μας βρίσκει διαφωνούντες στην Επιτροπή και μάλιστα έχουμε δει ότι τα κράτη-μέλη προσπαθούν να δαπανίσουν τα κονδύλια από το Ταμείο Ελληνικής μέσα στο χρόνο. Αν στο μέλλον μειώσουμε το χρονικό διάστημα από την καταστροφή μέχρι την ώρα της πληρωμής, η περίοδος εφαρμογής ενός έτους που επιτρέπει και αναδρομική χρηματοδότηση από την έναρξη της καταστροφής βραχύνεται, μειώνεται συνολικά και ίσως είναι λογικό να παρατείνουμε αυτή τη, αυτό το χρονικό διάστημα στο 1,5 χρόνο, 18 μήνες. Δεν διαφωνούμε. Αναφέρθηκε και η τεχνική βοήθεια. 2% τεχνική βοήθεια. Τώρα ο κανονισμός δεν προβλέπει τεχνική βοήθεια γιατί θεωρήθηκε ότι θα είναι σημαντικό να στηρίζουμε ε, επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης και όχι διοικητικές, όχι τις διοικήσεις. Το σύνολο λοιπόν των κονδυλίων του Ταμείου πηγαίνει σε επιχειρήσεις και όχι στην υποστήριξη των διοικήσεων ώστε να διαχειριστούν τα κονδύλια του Ταμείου. Αν θεωρηθεί ότι τα κράτη-μέλη όντως έχουν σοβαρές δυσκολίες και δεν μπορούν να εφαρμόσουν σωστά ε, χωρίς τεχνική βοήθεια τις προβλέψεις του Ταμείου θα το συζητήσουμε. Αλλά δεν έχει νόημα νομίζουμε να περιορίσουμε. Ε, νομίζουμε ότι ε, καλό θα ήταν να ε, μείνουμε στις περιοχές που καλύπτει το Ταμείο. Ευχαριστώ. Δηλαδή η τεχνική βοήθεια αναφέρεται και στους εμπειρογνώμονες γιατί μιλήσατε για διοικητικές δυνατότητες αλλά η ερώτηση του Νίκο, αφορούσε και τους εμπειρογνώμονες που θα μπορούσαν ίσως να κάνουν μια εκτίμηση επαγγελματικά και γρήγορα της ζημιάς, της καταστροφής. Εκ πείρας θα έλεγα ότι αυτό δεν δημιούργησε ποτέ δυσκολίες και υπήρξαν περιπτώσεις όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε ειδικού για να εκτιμήσουν ε, στην Λάκουιλα για παράδειγμα τις ζημιές που έγιναν. Και δεν ε, αντιληφθήκαμε ότι δημιουργήθηκαν από εκεί κάποιες ε, χρηματοδοτικές δυσκολίες. Αν κάποια μέλη ζητήσουν τεχνική βοήθεια, σκέφτονται ως επιτοπλίστων τη βοήθεια κάλυψης του διοικητικού κόστους υλοποίησης ή άσκησης του έργου ελέγχου και δεν ξέρω αν θα πρέπει να μπει σε, τέτοιες, σε τέτοιους τομείς στο Ταμείο ή σε επιχειρήσεις όπου υπάρχει άμεσο όφελος. Ο Λάμπερτ Βανίστελ Ρόι, κ. Βλάσα και μετά η σε επιχειρησεις οπου υπαρχει αμεσο οφελος ο λαμπερτ βανιστελ ροι ο βλασα και μετα Η συγγήτρια στο τέλος για να συνοψίσει, να ανακεφαλαιώσει. Θα είμαι, πολύ σύντομος. Αν ακούσετε όλες αυτές τις παρατηρήσεις, συνειδητοποιείτε ότι το όλο έργο δεν είναι καθόλου εύκολο. Υπάρχουν ε, όντως πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας που έχουν να κάνουν με τον κανονισμό αυτό καθ' αυτό αλλά και που σχετίζονται και με τους υπόλοιπους κανονισμούς που θα ισχύουν τα υπόλοιπα 7 χρόνια όσον αφορά τα υπόλοιπα ταμεία. Ας στηρίξουμε λοιπόν την εισηγήτριά μας. Βλέπουμε ότι Μπορούμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, αλλά δεν υπάρχει κανένα εχέγγυο, καμία απολύτω εγγύηση. Αν συνεχίσουμε να εργαζόμαστε όπω εργαζόμαστε μέχρι τώρα, δεν νομίζω ότι πρόκειται να λειτουργήσει το σύστημα, ιδίω στη συνεργασία που πρέπει να έχουμε με το Συμβούλιο. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, η Επιτροπή μα θα πρέπει ξεκάθαρα να πει ότι πρέπει να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα αυτό, η πρόταση αυτή, στην τρέχουσα νομοθετική ε, θητεία και ότι θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες συζητήσεις, ακόμα και τριμερείς διάλογοι για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Διαφορετικά πολύ φοβάμαι ότι θα μπούμε στο Φεβρουάριο, το Μάρτιο, θα πιέζει μετά πάρα πολύ ο χρόνος και οι περισσότεροι βουλευτές στη συνέχεια θα ασχολούνται περισσότερο με την ε, προκλογική τους εκστρατεία. Ενδεχομένω να πρέπει να στείλουμε και μια επιστολή και απευθύνομαι στην Πρόεδρο τώρα, προκειμένου να πείσουμε και το Συμβούλιο να συνεργαστεί μαζί μας πάρα πολύ έντονα και πολύ γρήγορα Ξέρετε ότι οι ειδικέ περιπτώσει χρειάζονται και ειδική αντιμετώπιση και νομίζω ότι ακριβώ αυτό ισχύει σε τη δική μα την περίπτωση. Ευχαριστούμε πολύ, Όλτζιχ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δράτω με τις ευκαιρίες για να σα δώσω και κάποιε πληροφορίε. Σήμερα και αύριο η Επιτροπή των Περιφερειών θα συζητήσει την έκθεση του κυρίου Μπράντα όσον αφορά το Ταμείο Λεγγύη Ευρωπαϊκή Ένωση Και νομίζω ότι θα πρέπει και οι συζητήσει αυτέ να ληφθούν από εμά υπόψη. Θεωρώ ότι ε, οι απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ανταποκρίνονται και σε διάφορα σημεία τα οποία εντοπίζονται στην έκθεση αυτή. Πρέπει να σας πω επίσης ότι η έκθεση είναι πλέον διαθέσιμη. Ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχουν σχόλια, δίνω το λόγο στη Ρώσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να κάνω μια σύνοψη Σήμερα το απόγευμα στις 4 θα με έχει προσκαλέσει ο πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών και θα λάβω το λόγο στο πλαίσιο της συζήτησης του Ταμείου Συνοχής. Αυτό σας το λέω ενημερωτικά, θα σημειώσω και τα δικά του αιτήματα. Ήδη έχουμε τη θέση τους γραπτός και κινείται προς την δική μας κατεύθυνση. Λοιπόν, περιφερειακές καταστροφές μέχρι τώρα ήταν κάτι το αόριστο, το αφηρημένο πιστεύω ότι στην πραγματικότητα, σύμφωνα με το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σημαντικότερο είναι να εφαρμόζεται η αρχή της αλληλεγγύης και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να βοηθήσει αυτές τις περιφέρειες. Τώρα τι γίνεται, ε, η συνδρομή δίδεται με βάση τον προϋπολογισμό και αν πληρεί τις ε, προϋποθέσεις των καταστροφών κλπ, ε, η χορήγηση βοήθειας γίνεται με βάση τον προπολογισμό και όχι τόσο πολύ με βάση την αρχή της ε, αλληλεγγύη. Αυτό είναι μια αυτοκριτική. Τώρα, εμείς θα προτείνουμε το 1% και στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου θα δούμε αν θα μείνουμε στο 1% ή, στο 1,5, ή θα πάμε στο 1,5%. Εμείς προτείνουμε 1% για να ε, μείνουμε πιο πιστοί στη συνθήκη σε ό,τι αφορά την ευθύνη των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, αντιμετώπιση τέτοιου είδους κρίσεων. Η Επιτροπή των Περιφερειών ζητάει επίσης 1%. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα της ξηρασίας που θα συμπεριληφθεί. Το ζήτησε και η Budget και η Επιτροπή των Περιφερειών. Και η σε τέτοιου είδου καταστροφέ όπω και στι πλημμύρε ε, θα πρέπει να υπάρχουν ειδικά μέτρα. Σε ό,τι αφορά την τεχνική σύνδρομη, η Επιτροπή των Περιφερειών είναι ομόφωνη για αυτό το θέμα. Γιατί πολλέ ε, περιφέρειε δεν έχουν, δεν διαθέτουν επαρκή εμπειρογνώμονε για να υποβάλουν φάκελο. Προφανώς το μεγαλύτερο κομμάτι των κονδυλίων θα πρέπει να έχει ως ε, σκοπό ε, την αποκατάσταση. Όμως για την υποβολή των ε, φακέλων χρειάζονται βοήθεια πολλές περιφέρειες διότι δεν έχουν δικό τους προσωπικό. Τώρα σε ό,τι αφορά τις υποδομές. Όπως είπε και η Επιτροπή των Περιφερειών θα προτείνουμε και εμείς το εξής. Πολλές φορές όταν υπάρχει μια καταστροφή αλλάζουν θέση υποδομές. Αν έχει περάσει για παράδειγμα ένας ανεμοστρόβιλος και καταστρέψει μια γέφυρα, μπορεί η γέφυρα να χρειαστεί να μετακομίσει αλλού. Σε ό,τι αφορά τις προκαταβολές, συμφωνώ με την budget. Να δούμε αν μπορούμε να λύσουμε το νομικό πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των 10 εβδομάδων, θα παρατείνουμε, θα ζητήσουμε παράταση αυτής της προθεσμίας, το ζήτησε και η Επιτροπή των Περιφερειών. Θέλουμε οι περιφέρειες να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία, χωρίς βέβαια να υπερβάλλουμε. 18 μήνες. Θα περάσουμε από τον ένα χρόνο στους 18 μήνες για την απορρόφηση. ναι νομίζω θα υπάρξει πρόβλημα εκεί. Σε ό,τι αφορά τις ΝΑΤΣ 2. Αυτό που ζητά η Επιτροπή των Περιφερειών είναι το εξής. Αν η καταστροφή λάβει χώρα σε περιφέρειες μικρότερες των ΝΑΤΣ 2 αλλά το σύνολο αυτών των περιφερειών να φτάνει σε πληθυσμό μια περιφέρεια να τις δύο, τότε να μπορούν να συμπεριληφθούν. Μετά, το θέμα της πρόληψης η Κομισιόν ε, υποτύπων εκ των προτέρων αιρεσιμότητας επιβάλλει συγκεκριμένες απαιτήσεις ό,τι αφορά τα μέτρα πρόληψης. Ε, η Επιτροπή των Περιφερειών ε, αμβλύνει αυτές τις ε, ε, ε, απαιτήσει ε, και εμείς θα κινηθούμε προς μια παρόμοια κατεύθυνση. Ασφαλώς και υπάρχει ένας κανονισμός οπότε το Συμβούλιο δεν βιάζεται, αλλά θα έπρεπε να προσπαθήσει να, και το Συμβουλίο να βελτιώσει το σύστημα γιατί το σύστημα αυτό μπορεί να βελτιωθεί και μάλιστα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για όλες τις τροπολογίες τις οποίες θα υποβάλλετε για να βελτιώσουμε το κείμενο. Ε, πιστεύω ότι θα φτάσουμε συμφωνία. Από την άλλη μεριά συμφωνώ και με τον κ. Βανίστερ Ρόι. Θα πρέπει να προλάβουμε πριν λήξει η θητεία μας. Ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται να αποφασίσουμε τίποτα σήμερα. Το χρονοδιάγραμμα ε, είναι το 18 Δεκεμβρίου παρουσίαση της έκθεσης, προθεσμία ε, για τις τροπολογίες και μέχρι τις 6 ε, Ιανουαρίου και ψηφοφορία 23 Ιανουαρίου. 23 Ιανουαρίου επίσης θα γίνει και μια δημόσια ακρόαση για το Ταμείο Συνοχής. Στις 23 έχουμε και συνάντηση με την Ελληνική Προεδρία. Θα ήθελα λοιπόν να σας προτείνω να κάνετε σαφές στην Προεδρία πόσο σημαντική είναι η έκθεση αυτή για μας και ότι θα πρέπει από κοινού να προσπαθήσουμε να κλείσουμε το ζήτημα αυτό κατά τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας. Αν αυτό δεν γίνει κατορθωτό, ο Μιγγέλ μου λέει ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να γίνει ψηφοφορία της για πρώτη ανάγνωση τον Απρίλιο και ενδεχομένως το νέο κοινοβούλιο που θα προκύψει ε, αποφασίσει να συνεχίσει από εκεί και να μην ξαναρχίσει από την αρχή. Υπάρχει μια τέτοια περίπτωση. Βέβαια το νέο κοινοβούλιο θα αποφασίσει, θα το δούμε. Θα συνεργαστούμε όμως με την Προεδρία στο μέτρο του δυνατού για να δούμε τι είναι κατορθωτό και τι όχι. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, ευχαριστώ για την Κομισιόν και περνάμε στις ψηφοφορίες. Να σας ενημερώσω ότι υπάρχει μια πρόταση αλλαγής ημερησίας διάταξης από το ΕΛΚ. Θέλετε να μας την παρουσιάσετε. Δεν έχουν έρθει όλοι για την ψηφοφορία ακόμα, οπότε να χρησιμοποιήσω το χρόνο που για να ζητήσω το εξής. Θέλω να μην ψηφίσουμε σήμερα την έκθεση Βόγκαν Οι συμβαστικές προτάσεις έφτασαν καθυστερημένα και για δύο από αυτές έχω κάποια ερωτηματικά. Μπορούμε να ψηφίσουμε στις 18 Δεκεμβρίου, αν κάτι τέτοιο είναι δυνατό. Θα ήθελα μια αναβολή αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Πρόεδρε, μπορείτε να ρωτήσετε τις υπόλοιπες ομάδες. Δεν θέλω να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες τώρα. Υπάρχει μια πρόταση λοιπόν να μην προβούμε στην ψηφοφορία της έκθεσης Βόγαν. Υπάρχει κανείς ε, που να διαφωνεί. Διαφωνεί κανείς, όχι. Ωραία. Η έκθεση Βόγκαν θα ψηφιστεί στην συνάντησή μας τον Δεκέμβρη. Οπότε ξεκινάμε την ψηφοφορία. Μπορούμε παρακαλώ να ελέγξουμε αν λειτουργεί σωστά το σύστημα ψηφοφορία, ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Αν άρχεται η ψηφοφορία, τεστ. Well, yeah. Oh. What a coordinator, yeah. Uh, dear colleagues, we have more... Έχουμε πιο πολλές κάρτες από ότι μέγιστο αριθμό Οπότε καλύτερα να ε, πατήσετε το κουμπάκι για να το λειτουργεί. Κλείνει η ψηφοφορία. Winkler, point 12 on our agenda. Σημείο 12. Έκθεση Winkler, ευφυής εξειδίκευση. Ψηφίζουμε τροπολογία 13. Υπάρχει μια προφορική ε, γλωσσική τροπολογία από τον εισηγητή. Όλοι συμφωνούν ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 15 και πάλι προφορική τροπολογία από τους σοσιαλιστές. Κανείς δεν διαφωνεί ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική πρόταση 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 με προφορική τροπολογία, κανείς δεν διαφωνεί με αυτήν. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, συμβαστική πρόταση 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παρακαλώ συγκεντρωθείτε και σηκώνετε τα χέρια σας. Τροπολογία 22 υπέρ. Ποιος είναι επικεφαλής στους σοσιαλιστές. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, συμβαστική πρόταση 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 37 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά τη 38 άρχεται ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 16 με 12. Τροπολογία 39 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε και την 39. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται 19 με 10. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 ε, υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 49 με προφορική σοφορία Υπάρχει κανείς που να διαφωνεί με την κατάθεσή της. Όχι. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά ελέγχουμε ηλεκτρονικά το 56 άρχεται η ψηφοφορία λίγη ψηφοφορία εγκρίνεται 19 υπέρ 9 κατά 60 υπέρ κατά Εποχές εγκρίνεται 17 συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά ελέγχουμε την 67 άρχεται η ψηφοφορία εγκρίνεται. 68 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 69 υπέρ, ελέγχουμε και την 69, άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας, εγκρίνεται, απορρίπτεται, συγγνώμη, απορρίπτεται, 18 κατά 12 υπέρ. Ε, συμβαστική πρόταση 1 για την ε, αιτιολογική έκθεση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 2, συμβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τσιμβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12. Με προφορική γλωσσική τροπολογία, διαφωνεί κανείς με την κατάθεσή της, όχι ψηφίζουμε υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο της ε, έκθεσης ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας. Δεν ξέρω γιατί, αλλά καλή έκθεση. Ε. Μερικές φορές όταν δεν είναι πριν αυτό το θέμα, δεν είναι καλές, αλλά συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Το 13 έχει ε, διαγραφεί τη μέση διάταξη, περνάμε στο 14, έκθεση Κάντενμπαχ. So, compromise... Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 και ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης ηλεκτρονικά τη ψηφοφορία. Πέρας. Ομόφωνα και αυτή εγκρίνεται. Εγώ όμως δεν ψήφισα, λέει πρόεδρος. Το ξέχασα. Μάλιστα, ολοκληρώσαμε λοιπόν τι ψηφοφορίε. Uh, uh, uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν πολλοί ακόμα στην αίθουσα και θα ήθελα να σας ε, ζητήσω και εφόσον έχουμε και λίγο περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας, και μόνο στις 10.30 μπορούμε να αναφερθούμε στην εξωτερική μελέτη, να περάσουμε ευθύ αμέσω στο σημείο 16 της ημερήσιας διάταξης ε, για τις Κανάριες νήσους είναι το θέμα εδώ πέρα. Ξέρετε ότι έχουμε μια απόφαση του Συμβουλίου για φορολογικέ απαλλαγέ ή ελαφρύνσει ε, του φόρου των προϊόντων που παράγονται τοπικά στι κανάριε νύσου. Δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε το ζήτημα αυτό. Πρέπει να εγκρίνουμε το νομικό πλαίσιο, το ρυθμιστικό πλαίσιο προκειμένου να μπορούν να ισχύουν τα μέτρα αυτά. Σας προτείνω λοιπόν να, να εγκρίνουμε με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χρησιμοποιώντας τον κανόνα 46 απλουστευμένη δηλαδή διαδικασία χωρίς τροπολογίες, άρθρο 46, χωρίς τροπολογίες. Νομίζω ότι ε, μπορεί να περάσει η απόφαση ε, κατά αυτόν τον τρόπο, εκτός και αν διαφωνούν πέντε μέλη της Επιτροπής μας. Είναι κάποιος κατά της πρότασης αυτής, ε, να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή το άρθρο 46. Αν συμφωνείτε, μπορούμε να αποφασίσουμε τώρα. Σας καλώ λοιπόν, μάλλον το ερώτημά μου, η έκκλησή μου είναι να αποδεκτείτε την απλουστευμένη διαδικασία του άρθρου 46 καθότι η απόφαση αυτή έχει ένα καθαρά τεχνικό χαρακτήρα και έναν επίγοντα χαρακτήρα, γιατί πρέπει να εγκρίνουμε στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου την απόφαση αυτή, προκειμένου να μπορούν τα προϊόντα από τις Κανάριες νήσους να χαίρουν αυτή τη φοροταπαλλαγή, γιατί ξέρετε ότι η φυστάμενη απόφαση θα εκπνεύσει τον Δεκέμβριο και θα βρεθούν οι Κανάριες νήσοι σε πολύ δύσκολη θέση. Αν δεν υπάρχει λοιπόν αντίδραση από τη δική σας την πλευρά, εγκρίνουμε την απόφαση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Νίκο, παρακαλώ, έχεις το λόγο. I don't hear you. Okay. As a group with um, Uh, Ω πολιτική ομάδα, με επιστολή του κυρίου Αλφόνση, του συντονιστή μας, ζητήσαμε από την Επιτροπή μας να κάνει μια ακρόαση όσον αφορά τα επιτεύγματα αλλά και τι αποτυχίε της πολιτική της ε, Τρόικα, όσον αφορά τις ε, πολιτικές ε, συνοχής. Ξέρετε ότι η ανάλογη διαδικασία έχει ξεκινήσει στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και θεωρώ ότι θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον και εμείς εδώ στη δική μας την Επιτροπή να έχουμε μια ακρόαση για τις επιπτώσεις της πολιτικής της Τρόικας όσον αφορά την πολιτική συνοχής και την περιφερειακή πολιτική. Κοιτάξτε, πρέπει με τους συντονιστές να ζητήσουμε το ζήτημα αυτό. Ελπίζω να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό το Δεκέμβριο και να λάβουμε μια απόφαση τότε το Δεκέμβριο. Αυτό που μπορώ να σας πω τώρα είναι ότι ε, παρακολουθώ εκ του Σύναγγη στη διαδικασία στην ΕΚΟΝ και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε μια ανάλογη συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη όμως τις ιδιαιτερότητες της δικής μας Επιτροπής. Δεν θα αποφανθούμε για την Τρόικα αυτή καθ' αυτή, αλλά περισσότερο για τις επιπτώσεις της πολιτικής της σε περιφερειακό επίπεδο. Δυστυχώς δεν είναι εδώ ο συντονιστής των σελιστών. Οι συντονιστές του ΕΛΚ από ό,τι φαίνεται δεν μας ακούν αυτή τη στιγμή. Διεξάγουν τη δική τους ιδιωτική συζήτηση. Θα ήθελα να αποφασίζαμε, αλλά το καλύτερο είναι να περιμένουμε να διεξαχθεί πρώτα η συνεδρίαση των συντονιστών. Δυστυχώ δεν με ακούν όμω αυτή τη στιγμή όπω βλέπετε. Πάντω στη συνεδρίαση των συντονιστών του Δεκεμβρίου θα συμπεριλάβουμε και αυτό το σημείο στη ημερήσια διάταξη. Ας περάσουμε τώρα στο σημείο 17 της ημερήσιας διάταξης, γιατί ο Γιώργος είναι εδώ μαζί μας. Υπάρχουν σκιώδεις εισηγητές για την απαλλαγή 2012. Δεν έχω λάβει σχετική πληροφορία. Γιώργο, έχεις το λόγο. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου μας δείχνει ότι το 2012 το ποσοστό σφάλματος στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής παρουσιάζει μία μικρή αύξηση σε σχέση με το 2011 από το 6% στο 6,8%. Ωστόσο αυτό που φαίνεται να μην γίνεται αντιληπτό ακόμα από αρκετού, αν ρίξετε μία ματιά στα δημοσιεύματα και σχετικές δηλώσεις, είναι το γεγονός ότι συχνά τα σφάλματα είναι διοικητικά και η ύπαρξη σφάλματος δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι οι πόροι έχουν χαθεί ή σπαταληθεί ή ότι έχει διαπραχθεί απάτη. Μπαίνοντα στην προεκλογική περίοδο θα συναντήσουμε αρκετέ προσπάθειε δραματοποίηση τη κατάσταση. Επειδή όμω οι αριθμοί δεν λένε ψέματα, χρησιμοποίησα στην έκθεσή μου τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μα για να θέσω την κατάσταση στην πραγματική τη διάσταση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη, στην πολιτική συνοχή στο 2012 οι παρατυπίε που κοινοποιήθηκαν ω δόλιες, ω fraud, αντιπροσωπεύουν το 0,42% των πληρωμών και οι συσσωρευτικές δημοσιονομικές διορθώσεις Cumulative Financial Corrections που πραγματοποιήθηκαν στο τέλος του 2012 για τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού ανάρχονται στο 0,2%. Φυσικά και υπάρχει περιθώριο για μεγαλύτερη βελτίωση. Στόχος μας οφείλει και πρέπει να είναι ένα μηδενικό ποσοστό σφάλματος και γι' αυτό θα πρέπει να καταβάλουμε περαιτέρω προσπάθειε και να μην επαναπαυθούμε μέχρι το να το πετύχουμε. Σε αυτή την προσπάθεια καλωσορίζω τι νέε ρυθμίσει που εισήχθηκαν στο Γενικό Οικονομισμό CPR για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, οι οποίες ελήφθησαν με τη διαδικασία της συναπόφασης, χάρη στις έντονες προσπάθειες που κατέβαλε η διαπραγματευτική μας ομάδα με επικεφαλής τον Λάμπερτ την Κωνστάζα και την πρόεδρό μας, αλλά και όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις. Οι κανονιστικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο Γενικό Κανονισμό, θα τις πω στα αγγλικά για διευκόλυνση, designations of Audit and Certifying Authorities, Accreditations of Audit Authorities, Audit Examination and Acceptance of Accounts, Financial Corrections and Net Financial Corrections, and proportional control στοχεύουν ακριβώς να συμβάλλουν στην περαιτέρω μείωση του επίπεδου του ποσοστού σφάλματος. Σας ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Ο Γιάνν Όλμπριχτ. Εγώ είμαι ο Σκιώδης για αυτήν την έκθεση για λογαριασμό του ΕΛΚ. Πρέπει νομίζω να γίνουν κάποιες σημαντικές παρατηρήσεις σε αυτό το στάδιο. Πάντα ε, ε, τίθεται ένα ερώτημα, τι σημαίνει ακριβώς απαλλαγή. Η απαλλαγή είναι η ανάλυση της έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου η απαλλαγή είναι το ερώτημα αν ταπανήθηκαν σωστά τα χρήματα ή όχι. Συχνά νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε την απαλλαγή ως καθαρή ανάλυση του κειμένου του ελεγκτικού συνεδρίου, παρόλο που γνωρίζουμε ότι το σύστημα των ελέγχων λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή το ελεγκτικό συνέδριο παίρνει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα και ελέγχει για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Αυτή είναι η ημερομηνία ελέγχου. Στο τέλος του έτους και μετά το, την παρέλευση του έτους γίνονται πολλές διορθώσεις. Οπότε η εικόνα διαφοροποιείται και δεν είναι εκείνη που ήταν τη μέρα του ελέγχου. Στο τέλος έχουμε μία πραγματικότητα η οποία διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια του έτους. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε την αναλλαγή ως αποτέλεσμα της ανάλυσης όλων των εγγράφων αυτό που κάνει εδώ η συγητής και στη Ρέντζη, δηλαδή πρώτα η έκθεση του ελεκτικού συνδρίου αλλά και η ε, αιτιολόγηση της έκθεσης της, του ελέγχου της Επιτροπής και ή επιθεωρήσεις που έγιναν μετά τους ελέγχους. Γιατί συχνά η επιθεωρήσεις που έγιναν μετά τους ελέγχους. Γιατί συχνά η εικόνα φαίνεται χειρότερη από ότι είναι στην πραγματικότητα. Ενώ ε, επικεντρώνουμε στην ημερομηνία ελέγχου, συχνά έχουμε πληροφορίες σχετικά με το ποσοστό των σφαλμάτων, αλλά αν συγκρίνουμε με τα πραγματικά δεδομένα διαφοροποιείται η κατάσταση. Ένα είναι αυτό λοιπόν. Δεύτερον, παρατηρούμε συνεχιζόμενη πρόοδο ενώ εντάσσομαι και άλλα μέσα στην πολιτική συνοχή. Όταν συγκρίνουμε τα δεδομένα των, διαφορετικών, των διαφόρων κρατών μελών σε διαφορετικές περιόδους, δεν ε, φαίνονται πολύ καθαρά. Αλλά νομίζω ότι τα μέσα αποσαφηνίζουν την κατάσταση και πρέπει να αναφερθεί. Επίσης, στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου σε τελευταία ανάλυση δεν έχουμε μόνο την ανάλυση του επίπεδου σφάλματος, αλλά έχουμε και την ανάλυση της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας των πολιτικών μέσα στο έτος. Αυτή είναι η ουσία της έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου και αυτό είναι μια ποιοτική αλλαγή στους ελέγχους. Επίσης, γιατί πολύ συχνά, και το έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, υπάρχουν προγράμματα και σχέδια τα οποία είναι απόλυτα ε, καθαρά, εις ό,τι αφορά το ποσοστό σφάλματος, αλλά είναι αναποτελεσματικά. Και αντίθετα υπάρχουν πολύ αποτελεσματικά έργα και προγράμματα τα οποία βαρύνονται από σφάλματα γιατί είναι καινούργια, είναι καινοτόμα και ακόμα δεν διαθέτουν την απαραίτητη πείρα. Τα σφάλματα λοιπόν είναι σημαντικά. Δεν σημαίνουν απάτη. Το σφάλμα μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας καινούργιας μεθόδου που δεν έχει πλήρως ελεγχθεί και νομίζω ότι πρέπει να συγκρίνουμε την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα με τα σφάλματα και μετά να αντλούμε συμπεράσματα για την ε, αποτελεσματικότητα της πολιτικής. Ο Μάρκος Πίπερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχω τη συνολική έκθεση για το Κοινοβούλιο και με που οι συνάδελφοι από την, Επιτροπή, την Περιφερειακή Επιτροπή δεν ε, επιμένουν στις βελτιώσεις που χρειάζονται. Αλλιώς θα είμαστε αναξιόπιστοι στην ευρωπαϊκή μας πολιτική. Καλύτερα να βάλουμε εμείς το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων παρά να το βάλουν οι ευρωσκεπτικιστές. Θυμίζω ότι είναι το τρίτο διαδοχικό έτος που έχουμε αύξηση του ποσοστού των σφαλμάτων. Αυτό δεν είναι καλό σημάδι. Επίσης το ελεγκτικό συνέδριο έχει ε, ελέγξει μόνο τέσσερις ελεγκτικές αρχές και όχι μάλιστα εθνικές ελεγκτικές αρχές από ε, χώρες όπου έχουν μεγάλα ποσοστά σφάλματος, αλλά άλλες χώρες και έτσι η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου είναι μάλλον αποδυναμωμένη. Και αν αυτή η αποδυναμωμένη έκθεση παρουσιάζει 6,8%, 6 ξέρω αυτό ήδη είναι ένα ανησυχητικό σημάδι. Και η περιφερειακή πολιτική πρέπει να ζητήσει τουλάχιστον βελτιώσεις. Δεν θα επικρίνω καθ' την περιφερειακή πολιτική, γιατί είμαστε περήφανοι για αυτά που καταφέραμε στην περιφερειακή πολιτική. Αλλά γεγονός παραμένει ότι οι συχνότητε των σφαλμάτων υπήρχαν στις ίδιες χώρες το 2000-2006, περίοδος που αξιολογείται, και για το 2007-2013 έχουμε τις πρώτες εκτιμήσεις επίσης και έχουμε πάλι σχεδόν τις ίδιες χώρες όπως και πριν που είχαν σφάλματα και έχουμε και καινούριες χώρες που με το σύστημα ελέγχου τους φαίνεται ότι έχουν προβλήματα και παρουσιάζουν κάποια ευάλωτα σημεία. Αυτό που είπε ο Γιώργος, ε, ότι γίνονται διορθώσεις, βεβαίως είναι σωστό αυτό, αλλά οι διορθώσεις μπορεί να πάρουν και δέκα 12 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν. Εν μέρη τα προγράμματα αντικαθίστανται από άλλα προγράμματα και ξανααντικαθίστανται από άλλα προγράμματα μέχρι να μπορέσουν να προωθηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια. Εν τω μεταξύ υπάρχει πρόβλημα από τον εθνικό προϋπολογισμό με την συνεχή επέκταση των προγραμμάτων και από το γεγονός ότι δεν αξιολογούνται με βάση τα ευρωπαϊκά κριτήρια. Τι ζημιά δημιουργείται έτσι από τον ενωσιακό, στον ενωσιακό προϋπολογισμό. Η ειλικρινής απάντηση πρέπει να είναι ότι χρειαζόμαστε κατεπηγόντως βελτιώσεις. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρενέσω να ε, επιδείξετε μεγαλύτερη τόλμη σε ό,τι αφορά την κριτική του συστήματος, χωρίς να θέλετε να το υπονομεύσετε. Βεβαίω θέλουμε να συνεχίσουμε την περιφερειακή μας πολιτική, αλλά αυτή τη ε, στιγμή έχω την εντύπωση ότι πάμε να κατευνάσουμε τα πράγματα. Και αυτό είναι κρίμα για το έργο της ε, περιφερειακή Επιτροπής. Ας είμαστε λίγο πιο θαραλέοι, ε, ζητώντας και πολιτικές συνέπειε από τα λάθη που έγιναν. Thank you very much. Any, any Ευχαριστούμε πολύ. Άλλες παρατηρήσεις. Γιάννης Νίλσεν. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Συμφωνώ ότι πρέπει ε, να ασχοληθούμε με την έκθεση αυτή πάρα πολύ σοβαρά και πρέπει τα συστήματά μας να αρχίσουν να λειτουργούν κάπως καλύτερα. Και ξέρετε ότι πρέπει να υπάρχει και απαραίτητη καταρτισμένη διοίκηση για να γίνει κάτι τέτοιο. Σε ορισμένε χώρε δεν συμβαίνει αυτό και θα πρέπει να γίνουν σε αυτές σημαντικές βελτιώσεις. Τώρα ποια είναι η εμπειρία από τη Σουηδία. Στη Σουηδία βλέπουμε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη διοικητική δομή η οποία ορθώνει κάποια εμπόδια για τις ε, περιφέρειες καθώς επίσης και τους επικεφαλείς των προγραμμάτων που θέλουν να χρησιμοποιήσουν κοινωτική χρηματοδότηση. Και πολλές φορές έχουμε και συγκρούσεις συμφερόντων, στις περιπτώσεις δηλαδή εκείνες όπου η Σουηδική διοίκηση εντοπίζει συγκρούσει συμφερόντων, ιδίως όσον αφορά τις συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Πιστεύω πάντως ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε κρατικά διοικητικά συστήματα τα οποία δεν θα δημιουργούν προβλήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι κρατικές διοικητικές δομές να διευκολύνουν τη χρησιμοποίηση της κοινωτικής χρηματοδότησης. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Λάμπερτ έχει το λόγο. Ε, προεκτείνοντας τα όσα είπε ο Γιάν, στην παράγραφο 5 της νομοδότησης γίνεται λόγος για τις επιπτώσεις των νέων κανονισμών. Και είναι αλήθεια όλα αυτά. Θα μπορούσαμε να είμαστε και λίγο πιο σαφείς, γιατί έχουμε πέντε ταμεία θα το δούμε και στο, στον τομέα της αλίας το ίδιο θέμα. Ε, και αν δούμε στην πράξη τι συμβαίνει, ε, στο παρελθόν κάναμε πολλούς διαφορετικούς υπολογισμούς για τη συνεισφορά των εταιριών σε είδος και έχουν γίνει πολλές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των ελέγχων. Τώρα εστιαζόμαστε πιο πολύ σε θεματικά πεδία, πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Έχει αλλάξει επίσης και η επικοινωνία ανάμεσα στις ε, διαχειριστικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε πιστεύω ότι αυτή η παράγραφος θα πρέπει να είναι πιο θετική έχουν γίνει πραγματικά πολλές απλοποιήσεις. Τόσο ότι αφορά αυτά που έλεγε ο Μάρκους για το πόσες χώρες ακολουθούν να έχουν προβλήματα ασφαλμάτων. Ασφαλώς και μας ανησυχεί, ανησυχεί την Επιτροπή μας. Αν δείτε τα νούμερα, δεν τα έχω μπροστά μου βέβαια, αλλά αν τα δείτε γνωρίζω ότι τα περισσότερα σφάλματα λαμβάνουν χώρες σε μικρό αριθμό χωρών, τις, στις ίδιες χώρες κάθε χρόνο. Θα πρέπει να έχουμε ένα ιδιαίτερο μηχανισμό να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ε, χώρες. Δεν είναι δυνατόν ε, τα σφάλματα γίνονται σε ένα μικρό αριθμό χωρών και να παίρνει όλες η μπόρα, να τις παίρνει όλες η μπόρα. Θα πρέπει να ε, είμαστε πιο αυστηροί με χώρες οι οποίες παρουσιάζουν υψηλό δείκτη σφαλμάτων και λιγότερο αυστηροί με χώρες οι οποίες ε, όλα τα τελευταία χρόνια δείχνουν να έχουν χαμηλό ποσοστό σφαλμάτων. Οπότε καταλαβαίνω τι λέμε εδώ, αλλά η εντύπωση μου είναι προσωπικά ότι Το ελεγκτικό συνέδριο μας ε, ε, ε, μάλλον βάζει στο ίδιο σακούλι όλο τον τομέα. Ο, όμως θα έπρεπε να γίνουν διακρίσεις. Υπάρχουν χώρες που έχουν ποσοστό το κάτω του 2%. Θα μπορούσαμε λοιπόν να δούμε πώς ε, ε, θα κάνουμε τα μέτρα αυτά να τα προσαρμόσουμε στην πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ε, και εγώ θέλω το λόγο τελικά. Να πω το εξής αφού κανείς άλλο θέλει το λόγο. Όλες αυτές οι δομές που ε, περιλαμβάνονται στο σημείο 5, δομές ελέγχου κατά βάση, είναι πολύ σημαντικές. όμως απλώς ε, ανακαλύπτουν και αποδεικνύουν τα σφάλματα δεν είναι προληπτικά. Δεν είναι προληπτική η δράση τους. Πιστεύουμε όμως ότι είναι πολύ σημαντική η νομική ασφάλεια. Γιατί πολύ συχνά οι κανόνες ερμηνεύονται διαφορετικά από την Κομισιόν, διαφορετικά από τον τελικό δικαιούχο, τελικά, διαφορετικά από τα κράτη-μέλη και το, συμβούλιο, το ε, ελεγκτικό συνέδριο έχει και τη δική του ερμηνεία. Και πολύ συχνά όλε αυτές οι ερμηνείε δεν συμπίπτουν. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό η Κομισιόν να εκδίδει κατευθυντήρες γραμμέ. Και βέβαια αν ξαναεκδοθούν κατευθείαν γραμμέ, θα είναι ένα πολυσέλιδο έγγραφο, πολύ περισσότερο από ό,τι το παρελθόν, οπότε δεν ξέρω αν θα βοηθούσε. Αλλά η βελτίωση της νομοθεσίας ε, για την εξασφάλιση της διαφάνειας, της νομικής ασφάλειας, της ε, σαφήνειας, είναι απολύτως απαραίτητη. Γιατί υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα στην πράξη, που πάρα πολλοί παρερμηνεύουν την νομοθεσία χωρίς κακή πρόθεση. Κάνουν κάτι και μετά οι ελεγκτές μετά μερικά χρόνια το ανακαλύπτουν, λένε ότι είναι παράτυπο και ιδιαίτερα δεδομένου ότι ε, ακόμα και οι εμπειρογνώμονε από διαφορετικά όργανα έχουν διαφορετική άποψη. Εμεί πολύ πρόσφατα είχαμε τρει νομικέ υπηρεσίε οι οποίοι είχαν τρει διαφορετικέ νομοδοτήσει, τρει διαφορετικέ νόμε. Ε, δεν το κατακρίνω, αυτή είναι όμω η πραγματικότητα. Το ίδια πραγματικότητα ε, διέπει και την ε, δράση όλων όσοι ε, υλοποιούν τα προγράμματα, ερμηνεύουν κάπως τους κανόνες και οι ελεγκτές τους ερμηνεύουν διαφορετικά. Ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς από την Κομισιόν ακόμα εδώ. Ε, αρχίσαμε νωρίς τη συζήτηση του θέματος. Θα ζητήσουμε από το Γιώργο να έρθει σε επαφή με την Κομισιόν ενδεχομένως, να δει αν ε, έχουν σχόλια. Και εσύ Μάρκος. Ε, ο Γιώργος σίγουρα θα είναι πολύ δεκτικός σε όλα αυτά τα σχόλια. Δεν ξέρω αν θες να πεις δύο λόγια για να κλείσουμε. Ναι, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ωραία. Θα είμαστε γενναιόδοροι προς εσένα. 17 Δεκεμβρίου η προθεσμία για τις τροπολογίες. Προς εσάς μάλλον όλους. Ε, υιοθέτηση από την Επιτροπή μας το Φεβρουάριο. Γιατί η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου θα υιοθετήσει δική της το Μάρτιο. Αν υπάρχουν αλλαγές θα σας ενημερώσουμε. Έχουμε χρόνο όμως για αυτή τη γνωμοδότηση. Ας κλείσουμε λοιπόν και αυτό το σημείο της μέσης διάταξης και ας περάσουμε στην εξ... στη μελέτη που ζητήσαμε Σημείο 15 της ημερησίας διάταξης. Εξωτερική μελέτη με θέμα διαδίκτυο, ψηφιακό θεματολόγιο και οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών της Ευρώπης. Θα δώσω το λόγο στους συντάκτες ή εν πάση περιπτώσει σε κάποιον που θα μιλήσει εκ μέρους των συντακτών. Η κυρία Ροζάνα Λιφόντ είναι εδώ από την ε, International Data Corporation που είχε αναλάβει αυτή τη μελέτη. Παρακαλώ. Um, Ευχαριστώ πολύ. Μ' ακούτε καλά. Καταρχήν, καλημέρα σε όλους. Επιτρέψτε μου να σας συστηθώ. Ίσως ε, είδατε κάπου την International Data Corporation και διαβάσατε ότι εργάζομαι για αυτούς, αλλά εγώ είμαι ανεξάρτητη σύμβουλος και συνεργάστηκα στα πλαίσια της μελέτης με το ΞΥΛ, που είναι το Κέντρο Βιομηχανικών Σπουδών ως ανεξάρτητη εξωτερική σύμβουλος και συνεργάζομαι με πολλές και διάφορες εταιρείες και δημοσίους φορείς. Το πεδίο εργασιών μου ε, αναφέρεται στον αντίκτυπο επιπτώσεις καινοτομιών, τις βιομηχανικές καινοτομίες και ειδικότερα τις ε, τεχνολογίες ε, πληροφορίας και επικοινωνίας ICT και τον αντίκτυπο που έχουν κοινωνικο-οικονομικά. Λοιπόν, να σας δείξω την ημερήσια διάταξη που σκιαγραφεί τα σημεία που θα παρουσιάσω. Πρώτα απ' όλα θα αναφερθώ στους στόχους της μελέτης, μετά θα σας πω κάποια πράγματα για τις ε, επόμενες τάσεις και προκλήσεις στον τομέα των ICTs, τεχνολογιών πληροφορίας επικοινωνίας. Μετά θα δούμε τα αναμενόμενα ωφέλη στην οικονομική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών όπως θα προκύπτουν από το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη. Στα πλαίσια των μελετών κάναμε και μελέτες περιπτώσεων μεμονωμένων για να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις των περιφερειακών πρωτοβουλειών και αυτό θα είναι το επόμενο σημείο. Ε, οι άλλες πτυχές που θα καλύψουμε αφορούν τις επιπτώσεις ε, στην περιφερειακή ανάπτυξη κάποιων οριζοντίων πρωτοβουλειών που είναι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο και τέλος ε, θα παρουσιάσουμε κάποια συμπεράσματα. Και τέλος, αν θέλετε, θα μου κάνετε ερωτήσεις. Νομίζω ότι υπάρχει χρόνος. Οι στόχοι της μελέτης και η προσέγγιση της μελέτης. Οι στόχη ήταν να καταλάβουμε ουσιαστικά κάτω από ποιες συνθήκες προϋποθέσεις το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη θα έχει επίπτωση στην οικονομική ανάπτυξη, μεγέθυνση και την κοινωνική ευημερία σε περιφερειακό επίπεδο. Το ψηφιακό θεματολόγιο περιλαμβάνει κάποιες πρωτοβουλίες ε, που ε, τις διαχειρίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άλλες πρωτοβουλίες τις διαχειρίζονται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Το άλλο βασικό ζήτημα ήταν να καταλάβουμε αν οι εθνικές και οι, αν σε οι πρωτοβουλίες σε νοσιακό και εθνικό επίπεδο είναι συμπληρωματικές. Αν λοιπόν αυτές οι πρωτοβουλίες σε νοσιακό και εθνικό επίπεδο είναι συμπληρωματικές προς τις περιφερειακές πρωτοβουλίες και τι αποτελέσματα δίνουν. Κάποιο τεχνικό πρόβλημα υπάρχει και δεν μπορεί η ε, κυρία να δει τις διαφάνειες. Τώρα, για τη μεθοδολογία χρησιμοποιήσαμε τη στατιστική ανάλυση και την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και όπως σας είπα κάναμε πολλές μελέτες περιπτώσεων και αναλύσαμε τα οριζόντια θέματα όπως τα λέμε, δηλαδή πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο. Δυσκολεύομαι λίγο που δεν βλέπω τις διαφάνειες. Τώρα, εις ό,τι αφορά τις τάσεις ε, των ICT, τεχνολογιών πληροφορίας ε, επικοινωνίας, ξέρουμε όλοι ότι σήμερα η τεχνολογία της πληροφορίας καθορίζεται από τις νεφέλες, τις και τα κινητά ευρυζωνικά δίκτυα και τη δημιουργία πολλών κινητών συσκευών και εφαρμογών και από τα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ στην κατά δηλαδή την οικονομία και την κοινωνία, σε δύο επίπεδα. Στην οικονομία έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο γιατί χρειαζόμαστε ε, υποδομές ε, προχωρημένες και η έξυπνη οικονομία στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών αλλάζει. Πρέπει λοιπόν οι διάφοροι συντελεστές παραγωγής να μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους. Επίσης ε, τα FEE συστήματα όλα είναι αλληλένδετα. Ίσως θα έχετε ακούσει ε, ε, τα διασυνδεδεμένα εμπορεύματα ή τη δικτύωση στο διαδίκτυο. Όλα αυτά επηρεάζουν πολύ τα κοινωνικο-οικονομικά θέματα και τις κοινωνικο-οικονομικές καινοτομίες, γιατί χρειαζόμαστε ε, περισσότερες δεξιότητες στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Χρειάζεται να αυξηθεί ο βαθμός του ψηφιακού γραμματισμού, γιατί χρειάζεται σε πολλές ιδιωτικές και δημόσιες υπηρεσίες. Είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να ε, διαθέτουν τον απαραίτητο ψηφιακό γραμματισμό για να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν όλες αυτές τις δυνατότητες. Επίσης οι πολίτες χρειάζονται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και ασφάλεια και οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις πρέπει επαρκώς να χρησιμοποιούνται. Αυτό δεν θα συμβαίνει αν δεν διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι όλα τα απαραίτητα μέσα για να προσλαμβάνουν αυτές τη, αυτά τα δεδομένα, αν δεν διαθέτουν δηλαδή τις σχετικές τεχνολογίες. Εσείς την έχετε λάβει την παρουσίασή μου νομίζω. Αυτές είναι οι τάσεις λοιπόν της τεχνολογίας που σας παρουσίασα ήδη. Αυτές οι τάσεις σημαίνουν ότι η καινοτομία της ψηφιακής οικονομίας ε, είναι αλληλένδετη οι καινοτομίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό η μία από την άλλη. Η παραγωγικότητα εργασίας, για παράδειγμα, εξαρτάται από τις κοινωνικές αλλαγές, εξαρτάται από την ικανότητα των ανθρώπων να τις χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες. Η καινοτομία στα προϊόντα και στις διαδικασίες εξαρτώνται για παράδειγμα από την διαθεσιμότητα δεξιοτήτων ICT. Αυτό είναι από τα πιο σημαντικά ε, ζητήματα σήμερα στην Ευρώπη. Όταν μιλάμε για τη βελτίωση της ψηφιακής καινοτομίας, διότι υπάρχει μια αντιστοιχία σημαντική μεταξύ προσφοράς και ζήτησης των ε, δεξιοτήτων αυτών στις τεχνολογίες πληροφορίας και ε, επικοινωνίας. Η γνώση αυτής της ε, αλληλεπίδρασης των παραγόντων δημιούργησε την ιδέα ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια πολιτική, ένα μέσον που θα στηρίζεται σε ένα λεγόμενο ενάρετο κύκλο, όχι φαύλο. Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη μάλιστα θα θέλει να ενεργοποιήσει ένα τέτοιο ενάρετο θα λέγαμε κύκλο με βάση την ιδέα ότι το διαλειτουργικό διαδίκτυο και οι υπηρεσίες χωρίς σύνορα αυξάνουν την ποσότητα περιεχομένων και υπηρεσιών. Και αν αυξάνεται ε, ο αριθμός περιεχομένων και υπηρεσιών, αυξάνεται και η ζήτηση για ταχαία δίκτυα. Και το βασικό είναι ότι οι επενδύσεις σε γρήγορα δίκτυα είναι βιώσιμες μόνο όταν υπάρχει υψηλή ζήτηση για τα δίκτυα αυτά. Αυτός ο λεγόμενος ενάρετος κύκλος λοιπόν πρέπει να δώσει κίνητρα για τη ζήτηση ώστε να γίνουν έπειτα ε, βιώσιμες και διατηρήσιμες επενδύσεις. Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη είναι ε, μία από τις 7 εμβληματικές πολιτικές της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και όπως σας είπα στηρίζεται στην ιδέα ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας ενάρετος κύκλος. Εκτός αυτού, οι ICT, οι τεχνολογίες της πληροφορίας επικοινωνίας, παίζουν σημαντικό ρόλο για την επίτευξη των άλλων εμβληματικών πολιτικών στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Α, συγγνώμη, μου φαίνεται ότι βιάστηκα. διότι οι ICTs είναι σημαντικές για την ε, πολιτική καινοτομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα επανεστιάσει την ε, έρευνα και την ανάπτυξη που είναι ε, το βασικό μέσο της Horizon 2020 για την επόμενη προγραμματική περίοδο Επίσης, οι ICTs είναι πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη οικονομίας ε, χαμηλής ε, χρήσης άνθρακα λόγω της χρήσης των έξυπνων δικτύων και των ε, υποδομών πληροφορίας και τέλος οι ICT είναι βασικές για τη δημιουργίες νέων ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας βέβαια. Τώρα πώς επηρεάζει το ψηφιακό θεματολόγιο την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη. Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη στηρίζεται σε 7 πυλώνες. Υπάρχει η ψηφιακή ενιαγορά, η διαλειτουργικότητα και τα πρότυπα, η εμπιστοσύνη, ασφάλεια κλπ. Και σε κάθε έναν από αυτούς τους πυλώνες υπάρχει μία σειρά δράσεων που πρέπει να αναλυφθούν και συνολικά οι δράσεις είναι 101. Αυτές οι δράσεις είναι νομοθετικά μέτρα ή επενδύσεις ή ήπια μέτρα. Και υποτίθεται ότι θα έχουν ένα αποτέλεσμα, έναν αντίκτυπο που θα καταστεί ορατός με βράχη και μέσο πρόθεσμα. Μέσο έως μακροπρόθεσμα θα υπάρχει αντίκτυπος στην περιφερειακή ανάπτυξη. τα αποτελέσματα που βλέπετε εδώ με χρώμα πορτοκαλί είναι κυκλικά αποτελέσματα και είναι τα αποτελέσματα που αναφερα, πριν από πέντε λεπτά. Είναι τα κυκλικά αποτελέσματα. Αν το ψηφιακό θεματολόγιο, για παράδειγμα, λειτουργεί σε επίπεδο δεξιοτήτων ICT, ο αντίκτυπος, το αποτέλεσμα, δεν θα περιορίζεται στην αγορά εργασίας μόνο, αλλά θα υπάρξουν ε, θα, ε, κι άλλα ωφέλη. Αύξηση της παραγωγικότητας μιας περιφέρειας, αύξηση της ζήτησης για επενδύσεις στα ευρυζωνικά ή τη χρήση ε, υπηρεσιών ηλεκτρονικών online. Οπότε υπάρχει μια κυκλικότητα του αντίκτυπου και αυτό σε τελευταία ανάλυση θα έχει αντίκτυπο στην οικονομική μεγέθυνση και την, οικονομική, και την κοινωνική ευημερία. Όπως είπαμε και πριν, αν οι δημόσιες υπηρεσίες ε, βελτιωθούν, εξοικονομείται χρήματα, χρόνο και μειώνονται οι αποκλεισμοί σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Τώρα, για να δούμε αν αληθεύουν όλα αυτά και αν όντω έτσι έχει το πράγμα, για να το δούμε αυτό, επιλέξαμε έναν αριθμό μελετών περιπτώσεων. Προσπαθώντας να αναλύσουμε τον αντίκτυπο αυτών των μελετών περιπτώσεων που επελέγησαν από όλη την Ευρώπη. Είχαμε στην Εσθονία, το Βερολίνο, την Ιταλία, στην Ούμπρια, στην Ανταλουσία, στη Λιθουανία, στην Κορνουάλη. και μια άλλη διαπεριφερειακή μελέτη περιπτώσεων. Οι μελέτες περιπτώσεων που επιλέξαμε επιλέγησαν και με βάση συγκεκριμένους τομείς. Δηλαδή ένας τομέας ήταν ηλεκτρονική υγεία, ένας άλλος είχε να κάνει με την ηλεκτρονική μάθηση, εκπαίδευση, ο άλλος είχε στόχο να στηρίξει την, ε, έγκριση, την ε, ε, ε υιοθέτηση ICT από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στην Ανταλουσία το, η μελέτη αφορούσε ε, στην μεγαλύτερη πρόσβαση στο, στα ευρυζωνικά δίκτυα. Πρόκειτο για μια επένδυση 150 εκατομμυρίων ευρώ εδώ σε μια περιφέρεια με πολύ χαμηλό ΑΕΠ. Τέλος κάναμε για, την, για το ψηφιακό γραμματισμό μια μελέτη περιπτώσεων και ε, το διαπεριφερειακό ήταν ένα πρόγραμμα για την ηλεκτρονική υγεία. Μελετήσαμε λοιπόν τον αντίκτυπο αυτών των ε, περιπτώσεων Προηγουμένως σας μίλησα για πιθανούς αντικτύπους ε, αποτελέσματα. Όλα αυτά τα εξετάσαμε. Κάθε μια από τις μελέτες περιπτώσεων έχουν αντίκτυπο, έχουν επιπτώσεις σε διάφορους τομείς. Εδώ στη διαφάνεια βλέπουμε τις διάφορες πρωτοβουλίες, δηλαδή μελέτες περιπτώσεων που αναλύσαμε και στις κάθετες στήλε έχουμε τα αποτελέσματα, πιθανά αποτελέσματα, την έκβαση. Κάναμε, πήραμε συνεντεύξεις και αναλύσαμε την εκτίμηση επιπτώσεων αυτών των πρωτοβουλειών και είδαμε ότι δεν έχουν αντίκτυπο μόνο στην περιοχή για την οποία σχεδιάστηκαν και όπου εφαρμόστηκαν, στην περιοχή από όπου άρχισαν. Για παράδειγμα, η ηλεκτρονική υγεία, η πρωτοβουλία αυτή για την Εσθονία, επηρέασε την αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα ε, την παροχή καινοτόμων δημοσίων υπηρεσιών και προϊόντων, την πρόσληψη ηλεκτρονικών υπηρεσιών, την ε, βελτιωμένη περιφερειακή εδαφική συνοχή, τη μείωση του κοινωνικού κόστους, τη βελτίωση του περιβάλλοντος και αλλού. Κάθε μια από αυτές τις πρωτοβουλίες ε, έχει λοιπόν πολύ μεγαλύτερα ωφέλη και θετικά αποτελέσματα από ένα. Και στο παράρτημα της μελέτης υπάρχουν λεπτομέρειες με στοιχεία για κάθε μια από αυτές τις μελέτες περιπτώσεων αν ενδιαφέρεστε να τα δείτε. Τώρα, η οριζόντια ανάλυση των μελετών ε, περιπτώσεων μας ε, δίνουν ε, κάποια διδάγματα. Καταρχήν υπάρχει μια ευρεία διάκριση μεταξύ των πρωτοβουλειών που αναλύσαμε, γιατί υπάρχουν ορισμένες που προωθούν την προσφορά των ICTs. Άλλες πρωτοβουλίες ε, προάγουν την ζήτηση για τις ICT και το διαδίκτυο. Άλλες επικεντρώνουν στην πρόσβαση και τη χρήση των ICTs. Άλλες ε, έχουν στόχο την αποτελεσματικότητα εναντί της ε, ε, ισότητας. Διαφέρουν δηλαδή οι πρωτοβουλίες μεταξύ τους. Όμως Παρ' όλα αυτά, οι πρωτοβουλίες που αφορούν την ισότητα έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε σχέση με την απόκριση δυνατοτήτων την κοινωνική συμμετοχή, επηρεάζουν όμως και συμβάλλουν σημαντικά έμεσα στην περιφερειακή ανάπτυξη λόγω της κυκλικής επίπτωσης αυτών των επενδύσεων. οι πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ε, αποδοτικότητα ε, ενεργοποιούν οικονομική μεγέθυνση αφού οι συντελεστές παραγωγής ε, είναι αποτελεσματικότεροι, πιο αποδοτικοί, αλλά συμβάλλουν και σε βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης. Αν ενεργοποιήσω με μία πρωτοβουλία, για παράδειγμα, για την εργασία, αυτή θα συμβάλλει στη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης και τη μείωση του κοινωνικού κόστους. Μπορεί επίσης να επιτύχει ψηφιακό γραμματισμό και να βελτιώσει τους στόχους ε, εδαφικής συνοχής. Συνολικά οι πρωτοβουλίες δείχνουν μικτά και γενικά ισορροπημένα αποτελέσματα, αντίκτυπο και ίσως αφορά την οικονομική μεγέθυνση και την ευημερία. παρά τους αρχικούς τους στόχους. Ε, τα δύο αποτελέσματα στην οικονομική μεγέθυνση και στην κοινωνική ευημερία και τα δύο φαίνονται και έχουν παρατηρηθεί σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή πάντα έχουν αυτά τα θετικά αποτελέσματα. Well, the Οι επόμενες δύο διαφάνειες σας δίνουν ένα παράδειγμα των δράσεων που χρηματοδοτούνται κυρίως από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κλπ. Για παράδειγμα, η περίπτωση Guadalinfo στην Ισπανία είναι project που έχει ε, στόχους ε, ισότητας, ε, αποφυγής αποκλεισμού κλπ. Έχει αποτελέσματα και στον ηλεκτρονικό αλφαβητισμό και στην συνοχή των τοπικών κοινοτήτων αποτελέσματα στην, στον ηλεκτρονικό αλφαβητισμό βελτίωσαν την ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου, ενώ από την άλλη μεριά η συνοχή της τοπικής κοινότητας επηρέασε την κοινωνική ευημερία. Ο αντίκτυπος που βλέπετε με κόκκινο χρώμα στη διαφάνεια ε, σε ό,τι αφορά το κάτω δεξί κουτάκι του οικονομικής ανάπτυξης είναι δύσκολο να ε, υπολογιστεί ήδη από τώρα για παράδειγμα ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. Όμως το αποτέλεσμα στην ε, αγορά εργασίας είναι ορατό αμέσως στην, από την τοπική διοίκηση. Η την προπόθεση βέβαια ότι οι συνθήκες ε, που επικρατούν είναι κατάλληλες. Για παράδειγμα, οι επενδύσεις που γίνονται πρέπει να είναι ο, η τοπική κοινότητα και οι επιχειρήσεις να είναι όριμες να δεχτούν αυτές τις επενδύσεις. Άλλο παράδειγμα, μάλλον όχι, οριζόντια ανάλυση των περιπτωσιολογικών μελετών έδειξε συγκεκριμένους ε, παράγοντες κλειδιά. Πολιτική ηγεσία σε περιφερειακό επίπεδο. Ένα νομικό περιβάλλον που να είναι έτοιμο και όριμο για την ανάπτυξη των επενδύσεων και η υπάρχουσα ...ανεπτυχμένη υποδομή ε, πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών. Άλλοι παράγοντες, επιπρόσθετα συμπληρωματικά προγράμματα στήριξης και μέτρα, καθώς επίσης και επενδύσεις και ε, μια νοοτροπία που είναι φιλική προς, την καινοτομία. Ε, Επίση, ένα άλλο παράγοντα ε, θετικό που ε, ε, συμβάλλει είναι η αποδοχή από, την, από το κοινό καθώς επίσης ε, και η συμμετοχή των εμπλεκομένων. Πολλές φορές ε, λαμβάνονται μέτρα ή αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες ε, τις οποίες δεν παρακολουθούν οι ενδιαφερόμενοι το κοινό. Χρειάζεται λίγο να τους δοθεί χρόνος για να τις κατανοήσουν και να τις συνοδεύσουν στην ανάπτυξή τους. Επίσης, εθνικές και υπερεθνικές πρωτοβουλίες έχουν ε, αντίκτυπο στην περιφερειακή ανάπτυξη. Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη έχει ε, λαμβάνει συγκεκριμένες ε, δράσεις ευθύνης των κρατών μελών και άλλες δράσεις ευθύνης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε το ερώτημα είναι πώς αυτές οι πρωτοβουλίες επηρεάζουν την περιφερειακή ανάπτυξη. Αναλύσαμε αυτό το, αυτή την πτυχή αναλύοντας μία υπερεθνική πρωτοβουλία, την ψηφιακή πανευρωπαϊκή υπηρεσία και ένα δεύτερο παράδειγμα που χρησιμοποίησαμε ήταν οι εθνικές πολιτικές ε, για ε, ικανότητες ε, ε, ICT. Τεχνολογία τη πληροφορία και των τηλεπικοινωνιών. Τα περάσω κατευθείαν στα συμπεράσματα. για να δώσουν αυτές τις πρωτοβουλίες ε, τα αναμενόμενα αποτελέσματα στην περιφερειακή ανάπτυξη υπάρχουν κάποιοι, κάποιες κάποιοι όροι. Ε, είναι για παράδειγμα, ότι θα πρέπει να αφαιρεθούν οποιαδήποτε εμπόδια πολιτιστικά, διοικητικά, ε, κανονιστικά, νομικά κλπ. Ο, επίσης, ο τοπικός πληθυσμός και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι έτοιμες ε, να υιοθετήσουν αυτές τις καινούριες τεχνολογικές λύσεις, γιατί αλλιώς οι επενδύσεις ε, δεν θα έχουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. η ε, πρωτοβουλία συνέδρου στην Ευρώπη θα είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την εφαρμογή των ε, στόχων του ψηφιακού θεματολογίου, αλλά ο συντονισμός και η χρηματοδότηση ε, είναι, δεν είναι επαρκείς συνθήκες, είναι αναγκαίες αλλά όχι επαρκές συνθήκες για την βιωσιμότητα των σχεδίων. Τώρα, πώς οι εθνικές ε, πρωτοβουλίες ε, στηρίζουν την ανάπτυξη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ε, η διασύνδεση ανάμεσα στα διάφο... στις δράσεις διαφόρων επίπεδων και τις της διακυβέρνησης στα διάφορα επίπεδα μπορεί να δώσει σημαντική ανάπτυξη. Πρωτοβουλίες από πάνω προς τα κάτω και project από κάτω προς τα πάνω θα πρέπει να συνδυαστούν ε, και να αναπτυχθούν συγχρόνως. Πολλές φορές όταν κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, οι δράσεις πολιτικής αποτυγχάνουν. Η εταιρική σχέση ιδιωτικού δημόσιου τομέα, η ΣΔΙΤ δηλαδή, είναι απολύτως απαραίτητη, απαραίτητες για το σχεδιασμό πολιτικών σε τοπικό επίπεδο προκειμένου να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα τοπικά ζητήματα και προκειμένου βέβαια να λάβουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Συμπεράσματα και συστάσεις. Πρέπει να εφαρμόζουμε όσο το περισσότερους τύπους μέτρων γιατί υπάρχει ένας κυκλικός χαρακτήρας, ε, μάλλον τα αποτελέσματα είναι κυκλικού χαρακτήρα. Σε, στον τομέα της ε, ψηφιακής καινοτομίας και ψηφιακής οικονομίας. Θα πρέπει τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας της πληροφορίας να ενταχθούν σε πιο πλατιές τιμικές στρατηγικές έτσι ώστε να συνοδευτούν από πρόσθετα μέτρα ε, που θα εστιάσουν στην αποτελεσματικότητα. Επίσης θα πρέπει να εντοπίσουμε το κατάλληλο μείγμα δημοκρατικής και ιδιωτικής στήριξης έτσι ώστε να πάρουμε τα κατάλληλα τοπικά μέτρα προσαρμοσμένα δηλαδή στις τοπικές πραγματικότητες. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι πληρούνται μια σειρά μια σειρά προϋποθέσεων έτσι ώστε να τα μέτρα που θα ληφθούν, οι, που θα αναλυφθούν να απορροφηθούν σε τοπικό επίπεδο. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ψηφιακό χάσμα αρκετά μεγάλο το οποίο θα πρέπει εμείς να ε, ε, γεφυρώσουμε. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ε, η, η τοπική η πραγματικότητα είναι ο σύνδρομος ανάμεσα στις οριζόντες και τις κατακόρυφες εταιρικέ σχέσεις. Τέλος, ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη ε, σε αυτό το παράξενο σύστημα πολιτικής διακυβέρνησης που χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε περιφερειακές πολιτικές, έχουμε ε, εταιρικές σχέσεις μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που αναπτύσσονται στην ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, εδώ είναι το email μου. Είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Μπορεί να ξεκινήσει τώρα η συζήτηση ο Βίκτορ Μποστινάρου, ο πρώτος ομιλητή. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όντω, έρχεται την κατάλληλη στιγμή, θα έλεγα η μελέτη αυτή, έχοντας κατά νου όμω το όλο περιεχόμενο της μελέτης σας, θα ήθελα να πω καταρχά ότι είναι σαφές, τουλάχιστον επί του παρόντος, ότι οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών και ο σχετικό κλάδος δεν θα πρέπει να θεωρηθούν επανάκια για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Θυμάμαι πριν από μερικούς μήνες διάβασα στον οικονομίστα μία μελέτη της Diana Φαρούρ όπου έλεγε ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε μία μείωση του κλάδου ICT στα πλαίσια της παγκόσμιας οικονομίας και αυτή η μείωση θα οφείλεται στο ότι θα έχουμε πολλές σημαντικές νέες καινοτομίε οι οποίες όμως θα αρχίσουν να παρουσιάζουν πτωτική τάση και αυτές και έπειτα θα έχουμε και την όλη οικονομική και κοινωνική κρίση. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο κλάδος των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών δεν μπορεί τελικά να προσφέρει ένα μεγάλο αριθμό θέσεων απασχόλησης και δεν συμβάλλει επίσης να διατηρηθούν κάποιες παλαιότερες θέσεις απασχόλησης, ενώ θα έπρεπε να έχουμε πολλές νέες δεξιότητες οι οποίες ανταποκρίνονται σε πολύ εξειδικευμένες θέσεις απασχόλησης. Θεωρώ λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Όσον αφορά επίσης το συνολικό αριθμό θέσεων απασχόλησης, ο κλάδος ICT θα εξακολουθεί να παραμένει σημαντικότατος παράγοντας, αλλά όχι καθοριστικός παράγοντας. Η οικονομική κρίση έχει καταδείξει ότι ε, ο κλάδος της πληροφορικής ή των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών δεν μπορεί να αντικαταστήσει εντελώς την βιομηχανία, τον κατασκευαστικό κλάδο ή τον κλάδο τον μετασχηματιστικό της παραγωγής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνδυάζονται και οι δύο αυτοί κλάδοι παράλληλα, τόσο βιομηχανία όσο και πληροφορική. Επίσης, σε σχέση πάντα με την οικονομική κρίση την οποία διανύουμε, θα ήθελα επίσης να έχουμε και μια πιο σφαιρική εικόνα των επιπτώσεων της πληροφορικής και των νέων αυτών τεχνολογιών στην Ευρώπη που πλήττεται από την κρίση. Εξαιτίας της λιτότητας έχουμε κάποιες δραματικές επιπτώσεις όπως η μείωση της πρόσβασης στα εκπαιδευτικά συστήματα, όχι μόνο στην Ήπεθρο και έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιοχές στην Ευρώπη αλλά και στα αστικά κέντρα. Επίσης, δεν υπάρχει επαρκής πρόσβαση στην εκπαίδευση, όπως σας είπα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχουμε και λιγότερες δεξιότητες, λιγότερες ικανότητες στον τομέα της ε, πληροφορικής και στον τομέα της χρήσης των τεχνολογιών, της πληροφορίας και των επικοινωνιών. Δεν καταφέρουν οι άνθρωποι να υποφεληθούν ε, από τα ευνοϊκά ωφέλη του κλάδου αυτού. Και αυτό μας οδηγεί τελικά σε ένα άλλο δράμα, σε μια άλλη μεγάλη καταστροφή, τον λεγόμενο ψηφιακό αναλφαβητισμό, που τον βλέπουμε έντονο σε πολλές ε, περιφερειακές περιοχές και ιδίως στην Ήπεθρο. Υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές στην Ευρώπη που αντιμετωπίζουν τις δραματικές αυτές συνέπειες του ψηφιακού αναρφαβητισμού και τις πιο δραματικές θα έλεγα ακόμα συνέπειες θα τις δούμε όταν θα αρχίσει να προκύπτει τελικά ένας κοινωνικός διαχωρισμός ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι θα είναι οι δήμονες, θα έχουν τις ικανότητες, τις δεξιότητες και πρόσβαση επομένως σε καλύτερες θέσεις εργασίας και πιο καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι δεν θα έχουν τις δεξιότητες αυτές και οι οποίοι τελικά θα παραγωνίζονται όλο και περισσότερο στα περιθώρια της κοινωνίας. Καταλαβαίνετε ότι η πρόκληση αυτή είναι τεράστια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, πρέπει να δούμε πώς ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίσει το ζήτημα των πιο ηλικιωμένων. Πώς μπορούν οι πιο ηλικιωμένοι να αποφεληθούν και αυτοί από την τεχνολογία ITC. Όχι μόνο για το ζήτημα της απασχόλησής τους και των αμοιβών τους, αλλά και για την ίδια την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Τελικά πάντα καταλήγουμε σε αυτό το ζήτημα του κοινωνικού αποκλεισμού και της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Ας μην ξεχνάμε όμως και κάτι ακόμα. Σας ευχαριστώ επίσης πάρα πολύ που αναφερθήκατε στη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Όντως, θεωρητικά τα πράγματα πρέπει να λειτουργούν θετικά και ξέρουμε ότι οι βασικοί πυλώνες ήδη αυτή τη στιγμή έχουν θεσπιστεί και ότι μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί τελικά η διευκόλυνση αυτή συνδέοντας την Ευρώπη. Δεν έχουμε όμως την απαραίτητη υποδομή ακόμα. Οι δυνατότητες μεταφοράς δεδομένων μας δίνουν τη δυνατότητα να μεταφέρουμε πάνω από 3 τεραμπάιτ, ποσό πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με το σημερινό 1,2 τεραμπάιτ δηλαδή μόνο. Η Ευρώπη όμως δεν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή όσον αφορά τον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Άλλες περιοχές του κόσμου βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Άλλες περιοχές του κόσμου είναι η κινητήρια δύναμη. Βλέπουμε ότι παράλληλα υπάρχουν ε, πάρα πολύ καταρτισμένοι μηχανικοί οι οποίοι φεύγουν από την Ευρώπη, η λεγόμενοι διαρροή εγκεφάλων. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι, ιδίω στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορία και επικοινωνιών, ψάχνουν πλέον δουλειά σε άλλε περιοχέ του κόσμου και όχι στην Ευρώπη. Επίση, η διευκόλυνση συνδέοντα την Ευρώπη θα αντιμετώπιζε θεωρητικά και τα προβλήματα τα ευρυζωνικά αν δημιουργηθούν οι νέες κατάλληλες προϋποθέσεις για την ευρυζωνική πρόσβαση, θα καταφέρνουμε σε όλη την επικράτεια των κρατών μελών να έχουμε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Έχουμε μάλιστα ένα δισεκατομμύριο χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο ψηφιακό χάσμα ανάμεσα σε εμά και σε αυτούς οι οποίοι επενδύουν, κάνουν σημαντικότερες επενδύσεις στις νέες αυτές τεχνολογίες. Επομένως, είτε θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια συνεκτική ψηφιακή πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα πρέπει κάθε χώρα να ακολουθήσει μια ξεχωριστή, μεμονωμένη πολιτική. Στη δική μου τη χώρα θα έλεγα ότι στον τομέα ICT τα πηγαίνουμε καλά. Είδαμε εκπληξή ότι η Ρουμανία στην παγκόσμια κατάρτιση όσον αφορά την πρόσβαση στο διαδίκτυο έρχεται δεύτερη. Πρόσβαση στο διαδίκτυο και πρόσβαση μάλιστα σε γρήγορο διαδίκτυο. Ουδέποτε όμως είχαμε μία συνεκτική εθνική πολιτική για τον τομέα αυτό. Ήτανε μάλλον χαοτική η πολιτική μας θα έλεγα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλήξει σε μία συνεκτική ψηφιακή πολιτική. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, πριν από δύο-τρεις εβδομάδες η όλη ανακοίνωση που ακούσαμε για το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη ήταν πολύ καλά από θεωρητική πλευρά, αλλά δεν είδαμε στην πράξη να έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Ο κύριο Βανίστερο έχει το λόγο. Θα ήθελα και εγώ να πω κάποια πράγματα. Στα πλαίσια τη επιτροπή μα έχουμε κάποιε τέτοιε σημαντικέ εξωτερικέ μελέτε και στη συνέχεια ακολουθούν εκθέσει από του συναδέλφου μα, οι οποίε καταλήγουν τελικά στην Ολομέλεια. Δεν προβλέπεται όμω μια έκθεση, έτσι δεν είναι, στην Επιτροπή μα. Ναι, ναι. είχαμε ολοκληρώσει μέχρι τον Ιούνιο τον προγραμματισμό για τις εκθέσεις. Έπρεπε κάποιος να έχει δηλώσει διαθεσιμότητα ή να έχει υποβάλει την υποψηφιότητά του μέχρι τον Ιούνιο. Ναι, όχι, σας λέω όμως τι γίνεται στην πράξη, τι διαπιστώνω εγώ αυτή τη στιγμή. Τι θα κάνουμε τελικά εμείς με την εξωτερική αυτή μελέτη. Έρχεται μια χρονική στιγμή όπου αρχίζει ο νέος προγραμματισμός και μια ερώτηση θα ήθελα να θέσω προς ε, την εισηγήτρια, τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουμε να συνδυάσουμε τις τεχνολογίες ICT, την θεματική συγκέντρωση την πολιτική συνοχής, πώς θα καταφέρουμε ουσιαστικά να συνδυάσουμε τις διαφορετικές αυτές δυνατότητες, γιατί βλέπω ότι υπάρχει ένας κατακαιρματισμός στις διάφορες περιφέρειες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε και το Περιφερειακό Ταμείο, το οποίο έχει θεματική ενότητα ICT, θα μπορούσαμε λοιπόν στο μεταγενέστερο στάδιο να δούμε αν μπορούμε να έχουμε και κάποια σχετικά προγράμματα ICT σε εθνικό επίπεδο. Σήμερα το πρωί λοιπόν συζητήσαμε για την ευφύ εξειδίκευση. Ουσιαστικά απευθυνόμαστε σε κάποιους παραδοσιακούς τομείς, αλλά το ζήτημα του ψηφιακού θεματολογίου είναι τελικά ένας οριζόντιος τομέας δεν αναφερόμαστε σε ένα συγκεκριμένο μόνο τομέα, αναφερόμαστε σε εφαρμογέ που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε πάρα πολλού διαφορετικού τομεί, στον τομέα τη εκπαίδευση για παράδειγμα, αλλά και σε πολλού άλλου. Επομένω, θα μπορούσαμε πραγματικά και με σοβαρότητα να ασχοληθούμε με τα ICT, στα εξειδικευμένα προγράμματα, τα θεματικά. Μέχρι στιγμής το ποσοστό ICT στα προγράμματα αυτά είναι πολύ μικρό. Τη στιγμή αυτή λοιπόν που έχουμε περισσότερα ακόμα χρήματα, περισσότερα κονδύλια για την περιφερειακή πολιτική και έχουμε και τη σύνδεση, τη διευκόλυνση συνδέοντα την Ευρώπη, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να επικεντρωθούμε περισσότερο στο ICT και τελικά βλέπουμε ότι έχουμε καταλήξει στο 1 δισεκατομμύριο μπορούμε να εντάξουμε το ICT και στην θεματική συγκέντρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αλλά αυτό όμως δεν αρκεί από μόνο του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να διασυνδέσουμε όλους αυτούς τους τομείς μεταξύ τους. Ενδεχομένως λοιπόν στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία, στα πλαίσια της Επιτροπής αυτής, να πρέπει να γίνει κάτι σχετικά. Αυτό ακριβώς είπε και ο μποστινάρο κύριος Μποστινάρου πριν από λίγο. Ευχαριστώ Λάμπερτο, Νίλσεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω σου ειδικά, οπότε παρακαλώ βάλτε τα ακουστικά σας. Συμφωνώ με τον κύριο Νίστελ Ρόι. Θα πρέπει να εμβαθύνουμε. Και συμφωνώ και με τον κύριο Μποστινάτσου. Ότι, τον κύριο Μποστινάρου, συγγνώμη, ότι υπάρχει ένα κοινωνικό πρόβλημα. Να πω όμως το εξής. Κοιτώντα τη Βόρεια Σουηδία και τη Βόρεια Φινλανδία, που είναι πολύ αεροκατοικημένε περιοχές, κάθε φορά που πηγαίνω εκεί, τους ρωτάω τι χρειάζεται για να δημιουργήσουμε ανάπτυξη και ε, θέσει εργασία εδώ πέρα και μου λένε πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες. Αυτό μου λένε ως νούμερο ένα και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Πρόσβαση σε γρήγορο ίντερνετ. Έχουν έρθει μηχανικοί από τη Γερμανία στη Βόρεια Σουηδία, ε, Ολλανδοί που, συγγραφείς που ζουν εκεί, Και μόλις βγουν από τις μεγάλες πόλεις και χρειαστεί να δουλέψουν εκεί, αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Πολύ δε περισσότερο αν έχει κανείς και πελάτες εκεί. Οπότε η απάντηση που παίρνω πάντοτε είναι χρειαζόμαστε πρόσβαση σε γρήγορο ίντερνετ. κανείς εκεί δεν επενδύει τα δικά του χρήματα. Θα πρέπει το κράτος και οι τοπικές αρχές να κάνουν τις επενδύσεις. Και αυτό βέβαια μπορούμε να το ενθαρρύνουμε με χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία και το κάνουμε. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα δράσεων σε πολύ μικρές κοινότητες όπου έχουν εγκατασταθεί οπτικές σύνες, υπόγειες κλπ. Παρ' όλα αυτά απομένουν πολλά πράγματα να γίνουν. Ακόμα και σε τουριστικά μέρη που έχουν φιλοξενούμενους όλο το χρόνο. Όταν γεμίζουν αυτά τα μέρη κατά τη διάρκεια του χειμώνα για σκι κλπ. εκεί δεν τα καταφέρνουν. Μπορεί το υπόλοιπο χρόνο παρόλο που έχουν τουρισμό να τα καταφέρνουν. Όμω στου μήνε αιχμή μένουν πίσω. Τώρα δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να το ρυθμίσουμε φέτο ή να περιμένουμε την επόμενη θητεία. Ευχαριστώ, Γιάννη. Γιάνν Άλμπριχτ. Έχουμε 100% συμμετοχή των μελών στη συζήτηση. Εντυπωσιακό. Ε, άλλο η ποσότητα, άλλο η ποιότητα, λέει ο κ. Φανίστελ ε, δύο πράγματα με εντυπωσιάζουν εδώ. Πρώτον, το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού θυματολογίου. Ποιοτικές αλλαγές στις περιφέρειες. Είναι σαφές ότι οι ποιοτικές αλλαγές λαμβάνουν χώρα με την εφαρμογή θεματολογίου. Δεύτερον, η δισταγμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν συζητούσαμε τα διευθυντικά ταμεία. Να σας θυμίσω ότι ο Επίτροπος ήθελε απαγόρευση επενδύσεων ε, σε τεχνολογίες προφορίες ε, σε πολλές περιοχές της περιφέρειας της Ευρωπαϊκής ε, Δεν ήθελε τέτοιες επενδύσεις. Εμείς του είπαμε ότι η πρωτοβουλία συνόδας στην Ευρώπη ήταν πάρα πολύ σημαντική για μας. Ε, δεν παραπονιέμαι όμως. Το λέω απλώς ως παρατήρηση. Στην συζήτηση για το ψηφιακό θεματολόγιο ε, το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν οι κρατικές ενισχύσεις και οι ασαφείς κανόνες σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές, μάλλον τις κρατικές επενδύσεις στις υποδομές με ιδιώτες που θα τις διαχειρίζονται και θα τις εκμεταλλεύονται αργότερα. Και ένα, από τα εμπόδια στις ε, περαιτέρω επενδύσεις σε αυτές τις τεχνολογίες ήταν αυτό. Δηλαδή είναι αντιφατικό. Έχουμε ένα πολιτικό στόχο, το ψηφιακό θεματολόγιο κλπ. και από την άλλη μεριά έχουμε προβλήματα τα οποία, στις κρατικές ενισχύσεις τα οποία δεν βρίσκουν λύση. Μπορεί να βρήκαν, αλλά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων δεν φαινόταν να βρίσκουν λύσεις αυτά τα προβλήματα, τα προβλήματα των κρατικών ενισχύσεων. Και αυτό είναι καταστροφικό γιατί ένα από τα βασικά στοιχεία είναι το κατά πόσον οι τοπικές αρχές αποφασίζουν να κάνουν επενδύσεις για τέτοιου είδους τεχνολογίες ή αν θα πρέπει να το αφήσουν αφήσουν, αφήσουν αυτές τις επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα. Δεν ξέρω αν κανείς μπορεί να το απαντήσει τώρα, αλλά αυτό για μένα είναι ένα από τα βασικά προβλήματα του ψηφιακού θεματολογίου σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Κουρσκή. Θα μιλήσω πολωνικά. Βάλτε τα ακουστικά σας. Πιστεύω ότι το ψηφιακό θεματολόγιο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το θεματολόγιο στο οποίο οι τεχνολογίες αναπτύσσονται τόσο γρήγορα που καλό θα ήταν να γίνεται μια έκθεση σε τακτά διαστήματα που θα μας ενημερώνει για όλα αυτά. Είπατε κυρία Πρόεδρε ότι τον Ιούνιο κλείνει η προγραμματική περίοδος για τις προσφορές αυτές και συμφωνώ με όλους όσους είπαν ότι πρέπει να κάνουμε μια έκθεση με βάση αυτή τη μελέτη ίσως στις αρχές της επόμενης θητείας του Κοινοβουλίου και αυτό είναι σημαντικό για δύο βασικούς λόγους. Εμείς προφανώς επικεντρωνόμαστε σε κάποια τεχνικά θέματα όπως ας πούμε βριζονικό ίντερνετ, 5G, αλλά έχουμε και νομικά θέματα πριν από 1,5 χρόνο στην Πολωνία είχαμε μαζικές διαδηλώσεις εναντίον της ΑΚΤΑ που περιορίζει την πρόσβαση στο διαδικτυακό περιεχόμενο. Και είχαμε τις διαδηλώσεις γιατί υπάρχουν πολλοί που τα καταφέρνουν πολύ καλά, επαγγελματικά, βρίσκοντας ε, θέσεις εργασίας ή δημιουργώντας θέσεις εργασίας online και φοβήθηκαν ότι θα χάσουν αυτή την ευκαιρία να συνεχίσουν λόγω κάποιων νομικών προβλημάτων. Όταν μιλάμε για περιφερειακή ανάπτυξη βέβαια επικεντρώνουμε περισσότερο στα βασικά διαθεσιμότητα του διαδικτύου. Αλλά πρέπει να κάνουμε εκθεσή στην επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου. Αυτό θα ήταν καλή ιδέα με βάση όλα αυτά. Σας Θυμίζω ότι αυτό γίνεται μέσα από πολιτικές ομάδες και ελπίζω ότι θα βρεθεί μια πολιτική ομάδα που θα αναλάβει να κάνει μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Ο Γιώαχιμ Ζέλερ. Ευχαριστώ πολύ. Με προκάλεσε να λάβω το λόγο κύριε Σόλμπριχ για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή 100%. Μετά από αυτά που είπε, θα ήθελα και εγώ να πω ότι το ψηφιακό θεματολόγιο το κουβαλάμε από εδώ και από εκεί σαν ε, Άγιο Δισκοπότηρο της Εκκλησίας αλλά θα πρέπει να δημιουργήσουμε και ευκαιρίες για μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών. Ε, αναφερθήκαμε στη διευκόλυνση συνδέοντας, για τη, συνδέοντας την Ευρώπη. Ε, είχε προβλεφθεί δόθηκε ένα ποσό 10 ε, δις για αεροκατοικημένες περιοχές και οι εταιρείε κινητής τηλεφωνίας είχαν παρέμβει και είχαν πει ότι δεν πρέπει το κράτος να παρεμβαίνει και πολύ σε ιδιωτική, στην ιδιωτική επιχειρηματικότητα. Ε, τώρα η δικτύωση των αστικών περιοχών είναι καλή. Στο Βερολίνο, για παράδειγμα, έχουμε και πολλούς παρόχους στο διαδίκτυο, στη γεννητή τηλεφωνία, αλλά και εκεί κάποιες ε, περιφέρειες δεν είναι τόσο καλά συνδεδεμένες περιφέρειες των αστικών περιοχών, δεν έχουν τόσο καλή σύνδεση. Πάντως αυτοί που διαχειρίζονταν τα δίκτυα πλήρωναν πολύ για να, στο παρελθόν για να βελτιώσουν τα δίκτυα, κάνοντας ένα οικονομικό αγαθό. Εν τω μεταξύ είδαμε και τη δραστηριότητα των Κινέζων επενδυτών στην Ευρώπη. Εν τω μεταξύ ολόκληρα δίκτυα και δικτυακές δομές έχουν αγοραστεί από Κινέζους επενδυτές. Και τώρα ε, βλέπω ότι δραστηριοποιούνται πάρα πολύ στις καινούριες τεχνολογίες με συνεχείς προσκλήσεις σε εκδηλώσεις. εν ώψη και της προεκλογικής εκστρατείας και μετά τις μεγάλες μάχες για τα διαρθρωτικά ταμεία, πρέπει να φροντίσουμε και για την πρακτική εφαρμογή των προγραμμάτων ε, που χρηματοδοτούνται από τα ταμεία. Να δούμε αν ε, επιτυγχάνουν υψηλή προστιθέμενη αξία ή μήπως ε, θα πρέπει να υπόκεινται σε μια συνολικότερη στρατηγική ε, για την προστιθέμενη αξία στην Ευρώπη. Επίσης θα πρέπει να δούμε και την ε, εξασφάλιση της πρόσβασης ε, στα νέα μέσα και σε περιοχές άλλες από τις μεγαλοπόλεις και τους αστικούς χώρους όπου η δικτύωση δεν είναι πολύ μεγάλη. Κοντά στο Βερολίνο, σε ένα ομόσπονδο κρατήδιο, εις ό,τι αφορά την απορρόφηση των διαρθρωτικών κονδυλίων, στο παρελθόν παρουσίαζε κάποια ελλείμματα. Έγινε ένα προγραμματισμός και εντωμεταξύ έχουμε και περιοχές εκεί που δεν έχουν τόσο μεγάλο πληθυσμό και, είναι και υπάρχουν και πιο απομακρυσμένες περιοχές που όμως τώρα συνδέονται με τα διαρθρωτικά ταμεία και βοηθούνται. Ε, πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε και με τους μεγάλους επιχειρηματίες, με τους ε, ε, παρόχους των, των δικτύων, γιατί πολλές φορές η οικονομία λέει ότι κάποια προγράμματα δεν παρουσιάζουν οικονομικό ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν δημόσιες επενδύσεις, κονδύλια, να αναλάβει δηλαδή το δημόσιο, να καλύψει κάποιες ανάγκες. Επίσης ε, καλό θα ήταν η Κομισιόν να μην ε, μας ε, κατακλείσει με υπερβολικά πολλές διατάξεις και να γίνει βασιλικότερη του βασιλέως ή παπικότερη του Πάπα για να αναφερθώ και στον καινούριο Πάπα που είναι πιο φιλελεύθερος από τον προκάτοχό του. Έτσι πρέπει να κάνει και η Κομισιόν. Μου λένε... Οι πράσινοι μου είπαν ότι ο κύριος Αλφόνση θα υποβάλει την γνωμοδότησή του. Επομένως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την μελέτη αυτή προκειμένου να προσδώσουμε μια πιο έντονη εδαφική διάσταση. Να πούμε δηλαδή ότι συμπεριλαμβάνουμε και τον τομέα αυτό από τη Γενική Διεύθυνση τώρα Ρέτζι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να κάνω κάποιες παρατηρήσεις και να απαντήσω. Ε, πράγματι οι επενδύσεις ε, σε αυτές τις τεχνολογίες είναι η δεύτερη προτεραιότητά μας. Ε, είναι βασική οριζόντια τεχνολογία, ε, σημείο κλειδί για πολλές αδράσεις για τον τομέα των υπηρεσιών σε σύγκριση με τον ε, δευτερογενή τομέα, θέλω να σας πω το εξή. Ασφαλώς και ενθαρρύνουμε τη, χρήση αυτών των τεχνολογιών και των διαρροτικών ταμείων στην βιομηχανία. Στην ε, ε, μελέτη δίδεται έμφαση στην σχέση ζήτηση και προσφοράς κάτι που αντιμετωπίζεται σφαιρικά. Αυτό έχει σχέση με τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες και με τις ε, στατικές ηλεκτρονικές, ηλεκτρονικές στατικές ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά το θέμα των κρατικών ενισχύσεων, τα κράτη-μέλη προετοιμάζοντας αυτές τις στρατηγικές και οι περιφέρειες βοηθούν ε, η προετοιμασία των κρατών μελών βοηθάει στη δημιουργία των φακέλων. Γιατί στην ανάλυση προσφάσεις και ζήτησης μπορεί να εντοπιστούν αδυναμίες της αγοράς και γι' αυτό το λόγο μπορεί να είναι κάτι προετοιμασμένος για θέματα ε, κρατικών ενισχύσεων. Θα ήθελα επίσης να σχολιάσω την, το αποτέλεσμα της ε, περιπτωσιολογικής ανάλυσης. Θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον ότι τα αποτελέσματα ε, δεν ήταν ομοιόμορφα σε ό,τι αφορά την παραγωγικότητα. Προφανώς δεν είχαν όλα ως στόχο την βελτίωση της παραγωγικότητας και της ε, ανταγωνιστικότητας. Κάποιοι, κάποια είχαν στόχους ε, κοινωνικής συμπερίληψης. Όμως, αν συγκρίνουμε τα δύο σχέδια της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου που είχαν σχέση με την ευρυζωνικότητα, θα δούμε τα αποτέλεσματα διαφορετικά θα πρέπει να το δούμε καλύτερα. Επίσης, τα αποτελέσματα ηλεκτρονικής υγείας από ό,τι φαίνεται δεν είχαν αποτέλεσμα πάνω στην παραγωγικότητα, κάτι που είναι πολύ ανησυχητικό. Σε ό,τι αφορά τις συστάσεις και τα σχόλια που έκανε ο κ. Φανής για παράδειγμα, να καλωσορίσω το γεγονός ότι υπογραμμίζεται η στρατηγική προοπτική, δηλαδή η ένταξη των ε, μέτρων αυτών στις στρατηγικές και εγώ θα ήθελα να προσθέσουμε και η στρατηγική ICT θα πρέπει να ενταχθεί στη συνολική στρατηγική, στις συνολικές στρατηγικές ε, εφιούς εξειδίκευσης. Αυτή η στρατηγική αντίληψη των πραγμάτων είναι πολύ σημαντική. Και είναι και πολύ σημαντικό επίσης ε, να εξασφαλίσουμε το κατάλληλο μείγμα πολιτικών μείγμα πολιτικών, αλλά ταυτόχρονα να προσθέσω και κάτι ε, το οποίο έχει σχέση και με τον συντονισμό και το timing των διαφορετικών παρεμβάσεων. Έτσι ώστε όλες αυτές οι παρεμβάσεις ε, να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτό έχει σχέση και με τις κοινοτικέ επενδύσεις, όπως για παράδειγμα τις επενδύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος συνδοντας την Ευρώπη. Εμείς στη Ρίτζιο λέμε ότι όταν ένα κράτος μέλος θέλει την χρήση κοινωνικών ταμείων για ε, ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς θα πρέπει να εξετάζει τα ήδη υπάρχοντα συστήματα έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε τη διαλειτουργικότητα. Τελευταίο σχόλιο. Υπάρχουν πολλά προβλήματα με τα project ICT. Έχουν τις μικρότερες απορροφήσεις στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού. Αυτό οφείλεται μερικές φορές σε θέματα, προβλήματα κρατικών ισχύσεων, άλλες φορές οφείλεται στην πολυπλοκότητα των project αυτών. Εμείς εξετάσαμε το θέμα της ευρυζωνικότητας ε, και τα διάφορα μοντέλα επενδύσεων, ε, σχέσεων κυριότητας, και λοιπά, προκειμένου να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες που ενδιαφέρονται. Επίσης έχουμε δώσει κατευθείαν γραμμέ για τα project ηλεκτρονικού εμπορίου και, ε, και σε συνδυασμό με συναδέλφους σε άλλες υπηρεσίες της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο στη συντάκτρια της μελέτης να πω ότι όταν συγκρίνουμε project μην ξεχνάμε ότι ε, βρίσκονται σε, διαφορετικά, σε διαφορετικές φάσεις του κύκλου ζωής τους. Ε, γι' αυτό το λόγο ενδεχομένως τα αποτελέσματα τα βλέπουμε σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Από την δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, συνεπώς θα δώσω το λόγο στην, ε, στην συντάκτρια της μελέτης. Uh, θα προσπαθήσω να δώσω κάποιες απαντήσεις και αν ξεχάσω τίποτα θα μου πείτε. Καταρχήν συμφωνώ και εγώ με αυτό που λέτε ότι καμιά φορά όταν συγκρίνεται τα αποτελέσματα διαφορετικών επενδύσεων ε, στα πλαίσια διαφορετικών ε, προγραμμάτων και έργων αυτά δεν είναι συγκρίσιμα γιατί δεν υπάρχει ένα συγκριτικό σημείο αναφοράς αφού η διάρκεια ζωής της τεχνολογίας μπορεί να διαφέρει γιατί κάνετε επενδύσεις σε διαφορετικές τεχνολογίες, σε διαφορετικούς τομείς ή κάνετε μια επένδυση σε τομείς με κάποιες βασικές διαφορές στην οικονομική δομή τους. Οπότε οι συγκρίσεις δεν διευκολύνονται. και από άποψη μεθοδολογίας δεν είναι και σωστό να επιχειρούμε συγκρίσεις. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας κάθε φορά το σημείο αφετηρίας μας, πώς έγινε η επένδυση κλπ. Κάποιος είπε, υπό μορφή ερώτησης, ότι η καινοτομία στην ψηφιακή οικονομία δεν είναι πανάκια που θα λύσει τα όλα τα σημερινά προβλήματα. Βεβαίως, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια οι επενδύσεις και η ζήτηση στις τεχνολογίες πληροφορίας επικοινωνίας της ICT θα μειωθούν. κυρίως διότι η ICTs σήμερα είναι η τεχνολογία εκείνη που βοηθάει τις επιχειρήσεις να εξοικονομούν χρήμα. Κατά την κρίση είδαμε ότι το σκεπτικό των επενδύσεων μέσα στις επιχειρήσεις κύρια ε, ε, κύριο προσανατολισμό είχαν την εξοικονόμηση του χρήματος. Η τεχνολογία της πληροφορίας δεν μείωσε μειώθηκαν ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Διότι οι επιχειρηματίες συνεχίζουν να επενδύουν εκεί για να εξοικονομήσουν χρήμα. Επίσης δεν νομίζω ότι μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στη διαδικασία ψηφιοποίησης της οικονομίας που είναι μια γιατί αυτή είναι μια τεχνολογία που εξυπηρετεί πολλούς στόχους. Είναι συντελεστής παραγωγής πια. Έχει γίνει ένα συντελεστής που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Δεν μπορούμε πια να κάνουμε πίσω. Διότι όλοι έχουμε smartphone όλοι έχουμε εφαρμογές. Εγώ δεν νομίζω ότι θα μειώσουμε τις επενδύσεις επειδή θα αποφασίσουμε ότι οι νεφέλοι και οι υπηρεσίε νεφέλης δεν θα είναι ενδιαφέρουσες, δεν θα έχουν ενδιαφέρον. Έχουν ενδιαφέρον, διότι το μεγαλύτερο κομμάτι της ευρωπαϊκής οικονομίας στηρίζεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και εγώ η ίδια είμαι μια ανεξάρτητη εξωτερική σύμβουλος, μπορώ να συνεργάζομαι με πολλές εταιρείε που χρησιμοποιούν την θέλη και το, τη χρησιμοποιώ και εγώ από το γραφείο μου. Και ε, όλα αυτά τα χρησιμοποιούμε έτσι όπως αναπτύσσονται για να δουλεύουμε. Η τεχνολογία της πληροφορίας αλλάζει τον τρόπο παραγωγής μας, τον τρόπο ζωής μας, τον τρόπο εργασίας μας. Ε, η ψηφιακή οικονομία σίγουρα δεν θα ε, αντικαταστήσει τη βιομηχανική παραγωγή, συμφωνώ. Είναι μια τεχνολογία, δεν είναι κάτι άλλο. Αλλά αλλάζει τον τρόπο της παραγωγής και της βιομηχανικής παραγωγής. Και αυτό είναι θεμελιώδες. Και πρέπει πάντα να το έχουμε υπόψη μας. Και όλα αυτά θεμελιώνονται από το εξής. Κατά την οικονομική κρίση η αγορά εργασίας είχε τεράστια προβλήματα είχαμε σοβαρή ανεργία στην Ευρώπη. Αλλά πιστέψτε με, δεν έχω τα στατιστικά στοιχεία εδώ μαζί μου, αλλά μπορώ να σας τα στείλω αν θέλετε, που δείχνουν ότι η ζήτηση για δεξιότητες ICT αυξάνεται και οι επιχειρήσεις δεν ξέρουν πού να τις βρουν αυτές τις δεξιότητες. Γι' αυτό η εκπαίδευση πρέπει να αλλάξει. Γι' αυτό δεν μπορούμε να πάμε πίσω και να αντιστρέψουμε ε, την τάση αυτή. Το σημαντικό στο ψηφιακό θεματολόγιο είναι ότι είναι μία πολιτική οριζόντια, βεβαίως δίκιο έχετε που το λέτε αυτό, η οποία βοηθάει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων από κοινού. Πρέπει όλα να τα δούμε. Όταν αναπτύξαμε αυτές τις μελέτες των περιπτώσεων, ε, είδαμε ότι είναι πιο εύκολο να υπάρχουν αποτελέσματα όταν υπάρχουν πολιτικές που καταπιάνονται με διαφορετικές όψεις των ICT. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Κάποιος μάλιστα είπε εδώ ότι είναι πολύ σημαντικό να αναλύσουμε όλες αυτές τις πτυχές μέσα από το πρίσμα τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης. αλήθεια είναι και αυτό. Έχουμε πολλά παραδείγματα στην Ευρώπη. Στην ε, αρχή της περασμένης δεκαετίας θυμάμαι ότι είχα κάνει πολύ μεγάλες μελέτες και έργα και για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις υπηρεσίες, δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες. Και τότε έλεγαν διάφοροι, α, ε, έχουμε δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες, αλλά κανείς δεν τις χρησιμοποιεί. Δηλαδή η αξιοποίησή τους είναι πολύ περιορισμένη. Γιατί? Λόγω προβλήματος ε, ψηφιακού γραμματισμού. Να το θυμόμαστε αυτό. Στην επόμενη δεκαετία οι πιο ηλικιωμένοι θα είναι άνθρωποι που θα έχουν αρχίσει να δουλεύουν με τους υπολογιστές και τα λάπτοψ ο ψηφιακός διαχωρισμός από την άποψη δηλαδή του ψηφιακού γραμματισμού μειώνεται. Και ένας άλλος τρόπος για να το δούμε αυτό είναι να αναβαθμίσουμε την εκπαίδευση αρχίζοντας από τους μαθητές μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση τα πανεπιστήμια. Στην Ευρώπη το έχουν καταλάβει στα κράτη-μέλη αυτό το πρόβλημα ότι η εκπαίδευση πρέπει να αλλάξει την προσέγγιση της. Αντίστοιχα με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει και στην παραγωγή, τη βιομηχανική παραγωγή να αλλάξουν ε, παραγωγικές προσεγγίσεις και μεθόδους, γιατί κάποιος είπε ότι είναι ένα θέμα οργάνωσης ναι, είναι μια τεχνολογία πολλαπλών στόχων. Αν δείτε ας πούμε τον αντίκτυπο μιας ιδιωτικής επένδυσης στις ICT, ε, ο αντίκτυπος είναι καλός όταν ταυτόχρονα γίνεται και αναδιοργάνωση της εργασίας στους κόλπους μιας επιχείρησης. Το ίδιο ισχύει για όλα τα επίπεδα μιας εταιρείας ή στα πλαίσια της οργάνωσης μιας κοινωνίας ή στα πλαίσια της οργάνωσης μιας περιφέρειας. Προφανώς είναι και πολύ σύνθετο πρόβλημα αυτό, γιατί σημαίνει ότι ποτέ δεν μπορούμε να το δούμε με μονομένα και μονόπλευρα και Και αυτό έχει να κάνει με αυτή την κυκλικότητα ε, του αντίκτυπου που ανέφερα στην αρχή της ε, παρουσίασής μου. Νομίζω αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Λαφόντη. Πραγματικά εκπροσωπώντας και όλα τα μέλη της Επιτροπής θα ήθελα να πω ότι η μελέτη αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική για μας γιατί βλέπουμε επίσης όχι μόνο τις ευρωπαϊκές πολιτικές αλλά και τις εμβληματικές πρωτοβουλίες που έχουμε στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020 ιδίως για τις περιφέρειες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να εστιάσουμε στις πρωτοβουλίες αυτές και να καταφέρουμε να προσεγγίσουμε την ψηφιακή ατζέντα από την περιφερειακή και τοπική σκοπιά. Ήταν πολύ σημαντικό ότι καταφέραμε να δούμε συγκεκριμένε περιπτώσεις project τα οποία έχει αξιολογήσει και καταφέραμε και εμείς να καταλάβουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις τους. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την παρουσίαση αυτή. Ολοκληρώνεται και η συνεδρίασή μας. Θα έχουμε την στις 17 Δεκεμβρίου τη συνεδρίαση Reggie Κότερς. Um, Κοκτέιλ με συγχωρείτε για την, Reggie θα γίνει στις 17 Δεκεμβρίου και έχουμε ένα γεύμα εργασίας. Μέχρι τις 21 Νοεμβρίου πρέπει να πείτε αν θα συμμετάσχετε σε αυτό. Θα έχουμε το κοκτέιλ λοιπόν στις 17 Δεκεμβρίου και την επόμενη μέρα 18 Δεκεμβρίου θα έχουμε την τακτική μας συνεδρίαση εδώ στο Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ.